έγγραφο αυτό έγινε εφετηρία για περαιτέρω συζητήσεις. Έγιναν αρκετοί τριμερείς ε, διάλογοι με θετικό αποτέλεσμα και θα σας ενημερώσω τώρα σχετικά με τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά τη συνάντηση με Κομισιόν και Συμβούλιο. Ξεκινώντας λοιπόν, νομίζω πως μπορούμε όλοι να δεχτούμε με χαρά τη συμφωνία αυτή, η οποία θα έχει θετικές επιπτώσεις για την ε, φαρμακοβιομηχανία στα κρατη Θα δώσει σταθερότητα στους επενδυτές, αλλά και ασφάλεια δικαίου στην βιομηχανία σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή και τον ε, τρόπο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία. ιδιαίτερα για τα φάρμακα. Τα γενώσιμα και φάρμακα είναι πολύ σημαντικό να απολαμβάνουν προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως με την προϋπόθεση τα φάρμακα αυτά να εξάγονται σε τρίτες ε, χώρες. Εδώ ισχύει αυτόματα η περίοδος προστασίας 5 ετών. Τα γεννόσιμα φάρμακα αυτά μπορούν να, να παρασκευάζονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος κατά την ε, περίοδο προστασίας, όμως δεν είναι δυνατόν να πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το διάστημα των πέντε ετών. Μπορούν όμως να εξάγονται σε τρίτες χώρες. Αυτό θα δίνει προστασία στους ε, παρασκευαστές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως ε, πρόκειται για μεγάλη επιτυχία και προστιθέμενη αξία σε ό,τι αφορά τα γενώσιμα και τα βιοπαρεμφερή φάρμακα. Μετά, παραγωγή για αποθήκευση και για δημιουργία αποθεμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, οι συζητήσεις ήταν αρκετά έντονες. Καταλήξαμε σε συμφωνία για ε, μία περίοδο έξι μηνών. Σε ό,τι αφορά την ε, αποθήκευση πριν τη λήξη της ε, περίοδου προστασίας. Με το που παρέλθει η ημερομηνία λήξης της περίοδου προστασίας θα υπάρχει δυνατότητα να επανενεργοποιεί είτε η συμφωνία πολύ γρήγορα και οι παρασκευαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στην ε, αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γενώσιμα φάρμακα. Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις για τους παρασκευαστές γενώσιμων φαρμάκων, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν κοινοποίηση παραγωγής, η οποία θα κοινοποιείται και στον κάτοχο των ε, δικαιωμάτων αλλά και στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο θα γίνεται η Παρασκευή. Η κοινοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνεται μάλλον πρέπει να γίνεται το πολύ τρεις μήνες πριν την έναρξη της παραγωγής. Επίσης θα υπάρχει υποχρέωση σήμανσης των γενώσιμων φαρμάκων σύμφωνα με τις ε, προδιαγραφές και οι παρασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους ε, προμηθευτές για το ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου προστασίας ε, το φάρμακο αυτό μπορεί να εξαχθεί, δεν μπορεί όμως να απολυθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υπάρχουν σε ευδιάκριτο σημείο έτσι ώστε τα φάρμακα αυτά να μην πολλούνται εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά προς το παρόν. Να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές, ε, διότι η διαδικασία ήταν πάρα πολύ σύντομη, δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Καταφέραμε όμως να εργαστούμε ομαλά και αποτελεσματικά. Και θεωρώ πως η συμφωνία είναι καλή. Επίσης, θεωρώ πως η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να γίνει πράξη προτού τη λήξη της κοινοβουλευτικής ε, θητείας, διότι έτσι πιστεύω θα στεφτούν οι προσπάθειές μας με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόλκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θεωρώ και εγώ πως ε, το αποτέλεσμα στο τέλος ήταν ικανοποιητικό. Νομίζω πως η σκληρή δουλειά που έγινε εδώ στην Επιτροπή είχε αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση. Νομίζω πως καταφέραμε να περάσει η γραμμή μας. Δυστυχώς όμως μόνο για το διάστημα των έξι μηνών. Ε, υπάρχει μεγάλη απόκληση από την αρχική μας θέση των δύο ετών. Όμως ε, θεωρώ πως ε, παρόλα αυτά έχει γίνει το πρώτο βήμα για την ε, καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν πως η απόφαση είναι σωστή και πως χρειάζεται μία πολύ ισχυρή ρήτρα αναθεώρησης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά που έχουμε αποφασίσει θα εφαρμοστούν και θα ε, ωφελήσουν τα μέγιστα τους ε, ασθενείς. Στον ε, τριμερή διάλογο μάλιστα έγινε υπέρβαση κατά μία ώρα της προγραμματισμένης διάρκειας και αυτό γιατί κύριο μέλημά μας είναι η υγεία των ασθενών. Σας ευχαριστώ πολύ. κύριος Καφαντά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Διότι ο κύριος Ζεύκα και ο κύριος Μπόλκεν είπαν τα βασικά. Ήθελα μόνο ε, να πω τρία πράγματα εν συντομία. Ε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους μου τον κύριο Σεγητά, τον κύριο Γκράντες Πασκουάλ, κύριε Βίσκα, ε, Ζήφκα, μάλλον για την εξαιρετική ε, στάση του καρδιά και της διαπραγμάτευσης. Ε, με όλους, προσπάθησε να βρει ε, συμβαστικές λύσεις ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Ε, το δεύτερο είναι ότι βάζουμε τέλος σε αυτήν το μειονέκτημα το ανταγωνιστικό το οποίο ζούσαν πολλές επιχειρήσεις φαρμακευτικές και έρευνας στην Ευρώπη και βέβαια η προστασία της έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν πρέπει να υπάρξει εδώ μια ρογμή. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε αυτές τις εταιρείε ε, της επιχείρησης και για τα ζητήματα αυτά πνευματικής διοκτησίας. Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος συναδελφός το λόγο, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό της σημερινής διάταξης και να συνεχίσουμε με το σημείο 20 υποβολή αναφορά στην Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο. Το λόγο έχει ξανά ο κύριος Σβιεύκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα ψηφιακά εργαλεία λοιπόν και διαδικασίες στο εταιρικό δίκαιο. Εδώ γίνεται λόγος για την ε, επιγραμμική εγγραφή εταιριών και των θηγατρικών τους. Στόχος είναι να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες. Με το να συντομεύσουμε τη διαδικασία εγγραφής καταχώρησης και να ε, γίνει αυτή η διαδικασία πιο οικονομική. Τα ψηφιακά εργαλεία λοιπόν θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους, όχι μόνο για τις επιγραμμικές συναλλαγές, αλλά και για τις ε, διαδικασίες ε, καταχώρησης των εταιριών. Να τονίσω ότι πρόκειται για εργαλείο που θα χρησιμοποιείται προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά. Έγινε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων ε, κατά τη διάρκεια του τριμερού ε, διαλόγου, αλλά και στις ε, διάφορες τεχνικές συζητήσεις. Εκεί προσπαθήσαμε να εξετάσουμε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες. Καταφέραμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας χάρη στην εξαιρετική δουλειά όλων, ιδιαίτερα της ε, Ρουμανικής Προεδρίας και της Επιτρόπου Γιουρόβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το δικό μας επιτελείο, το επιτελείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να πω ότι στον τελευταίο τριμερή διάλογο ολοκληρώσαμε τις εργασίες στα τελευταία αναπομείναντα τεχνικά ζητήματα τα οποία απαιτούσαν κοινή συμφωνία όλων, οι οποίοι έπρεπε να είναι παρόντες στην διαδικασία. Η... Συζητήθηκε λοιπόν η περίοδος ε, διαρκείας της οδηγίας, η πρόσβαση στην πληροφορία, η χρήση των ψηφιακών εργαλείων και η τελική έγκριση του κειμένου ιδιαίτερα των σημείων εκείνων που αναφέρονται στην υποχρέωση φυσικής παρουσίας κατά τη διάρκεια της ε, εγγραφής. Φυσικά, φροντίσαμε να διατηρηθεί ε, το σκεπτικό της ε, επιγραμμικής δυνατότητας καταχώρησης μιας εταιρείας. Και επίσης επικεντρωθήκαμε τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο της εφαρμογής στις ε, ιδιωτικές επιχειρήσεις διότι προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις ε, ανάγκες των ε, κρατών μελών σε αυτό το στάδιο πάλι. Πρόκυψε ένα θέμα νομικού χαρακτήρα Πρόκειται για ένα παροχημένο εργαλείο, τουλάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια μορφή δηλαδή εταιρικής σχέσης η οποία δεν ε, υφίσταται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίοδος εφαρμογής της οδηγίας έχει οριστεί στα δύο έτη με πιθανή παράταση ενός ακόμα έτους εφόσον τα κράτη-μέλη το επιθυμούν. Εάν κάποιο κράτος μέλος ε, επιθυμεί λοιπόν να δοθεί παράταση στην εφαρμογή της οδηγίας, θα πρέπει να κοινοποιήσει την πρόθεσή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να την αιτιολογήσει. Τώρα ένα άλλο ζήτημα αρκετά πολύπλοκο είναι ότι για ορισμένους ανθρώπους ε, δεν θα προβλέπεται δυνατότητα συμμετοχής σε διοικητικές θέσεις σε ορισμένες εταιρείε. Αυτό γιατί είναι σημαντικό, ε, διότι όταν διοικεί σε μια εταιρεία πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν αντικρούμενα συμφέροντα. Αυτά ως προς την ε, δομή του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν θεσμεύθηκε να αναθεωρήσει την οδηγία μέσα σε έξι χρόνια μετά την ε, υιοθέτησή της. Καταφέραμε να μειώσουμε το χρονικό διάστημα αυτό, διότι αρχικά το σκεπτικό της Κομισιόν ήταν ε, να αναθεωρηθεί η οδηγία μετά από δέκα χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση στην πληροφορία και το μητρό μιας εταιρείας. Τα μετρό αυτά σε πολλές περιπτώσεις χειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες έτσι ώστε πρώτον ε, να, καλύ... πρώτον, ε, να καλύψουν το κόστος κατόπιν αμοιβής. Ήταν λοιπόν δύσκολο για εμάς να αξιολογήσουμε ε, το εάν οι πληροφορίες για μια εταιρεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμες δωρεάν για κάποιο τρίτο μέρος. Καταλήξαμε λοιπόν ε, τελικά σε μια λύση η οποία από τη μία προστατεύει τις ιδιωτικές οντότητες ε, οι οποίες έχουν μητρώα καταχώρηση εταιρεών, από την άλλη επιτρέπει διατροπώντας την πρόσβαση για σημαντικούς λόγους. Θα υπάρχουν και ορισμένες πληροφορίες οι οποίες δεν θα είναι προσβάσιμες και αυτές αφορούν τον αριθμό των εργαζομένων σε μια εταιρεία διότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αλλάζει από χρόνο σε χρόνο. Εάν θέλουμε λοιπόν να φαίνονται οι αλλαγές στον αριθμό των υπαλλήλων θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλες ε, παραμέτρους και αυτό είναι κάτι που θα κάνει πιο δύσκολη την αξιολόγηση γι' αυτό και το αποφύγαμε. Μετά οι πληροφορίες που θα διατίθενται θα αφορούν το νομικό καθεστώς μιας εταιρεία, Δηλαδή πότε έγινε η καταχώρηση, πότε αφαιρέθηκε μία εταιρεία από το Μητρό. Το ίδιο και για τις ε, θηγατρικές. Πότε δηλαδή έγινε η καταχώρηση μιας θηγατρικής. Επίσης, θα είναι διαθέσιμες πληροφορίες για τον ή τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν την εταιρεία στις επαφές της με άλλες οντότητες. Νομίζω λοιπόν πως καταφέραμε να επιτύχουμε μία ισορροπία η οποία είναι ικανοποιητική για όλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φυσική παρουσία ορισμένων ατόμων, προσπαθήσαμε να διατηρηθεί το ε, σκεπτικό της επιγραμμικής καταχώρησης μιας εταιρείας. Αλλά εάν υπάρχουν δυσκολίες στην ταυτοποίηση κατά την διάρκεια της επιγραμμικής καταχώρησης, χρησιμοποιούμε μία ε, αρχή σύμφωνα με την οποία το κράτος μέλος θα ζητήσει από τον ε, θα ζητήσει τη φυσική παρουσία του ετούντο. Τώρα, στις 14 Φεβρουαρίου, το Συμβούλιο δέχτηκε την ε, συμφωνία που επετεύχθη στον τριμερή διάλογο και τώρα περνάμε στα επόμενα βήματα προς την τελική έγκριση. Θέλαμε να ολοκληρώσουμε στην συνάντηση αυτή, σε εκείνον τον τριμερή διάλογο. Όμως για να βοηθήσω τον κύριο Γκούτελαντ ε, καταλήξαμε στο να ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Ελπίζω λοιπόν να φτάσουμε στο τέλος και να πέσει αυλαία εντό ε, της κοινοβουλευτικής ε, που διανύουμε στην Ολομέλεια του Απριλίου μαζί με την ε, ψηφοφορία για την έκθεση της κυρίας Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο τον λόγο. Η κυρία Γιούτελαντ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Νομίζω ότι είχαμε επικοδομητικές, ε, καλές συζητήσεις στον τριμερή διάλογο και φτάσαμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουμε αυτήν την εντολή από το Κοινοβούλιο και είχαμε τη δυνατότητα έτσι να είμαστε ισχυροί στον τρίλογο. Βεβαίως ήταν επικοδομητικός και ο εταίρος μας στο διάλογο αυτόν. Το Συμβούλιο από την αρχή ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ωφέλη της εσωτερικής αγοράς, να δημιουργήσουμε ένα καλό πεδίο ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Ε, θα φροντίσουμε λοιπόν να συμβεί αυτό στο μέλλον, να υπάρχουν όμω ταυτόχρονα και οι απαραίτητε δικλείδε ασφαλείας, έτσι ώστε ε, να μην ε, έχουμε αρνητικέ επιπτώσει στην εσωτερική αγορά από ασόβαρες επιχειρήσεις. Φτάσαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα νομίζω. και αυτή η νομοθεσία θα βελτιώσει τα πράγματα. Το εταιρικό δίκαιο βέβαια είναι ένα πακέτο και θα πρέπει να ψηφίσουμε από κοινού ε, για το επόμενο νομοθέτημα που θα συζητήσουμε σήμερα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν φαίνεται να θέλει κάποιος άλλος το λόγο για το θέμα αυτό, το 20 δηλαδή. Μπορούμε λοιπόν να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Μιας και δεν είναι εδώ ο εισηγητής για το σημείο 21 Εγκαθιστάτε την κυρία Ρέγνερ ε, Ναι ωραία πάμε στο σημείο 21 Έκθεση λοιπόν στην Επιτροπή για τις διασυνοριακές ε, ε συγκλήσεις, ε, συγχωνεύσεις και διαχωρισμούς Έχετε το λόγο Ναι θα ήθελα στο όνομα της Εύλιν Ρέγνερ να σα δώσω αναφορά. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι εδώ, μου έχει δώσει όμως κάποια στοιχεία για το τι συμβαίνει εκεί. Μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Γιούρη στις 6 Δεκεμβρίου πέρυσι, ε, η εντολή επιβεβαιώθηκε στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου με συντηρητική πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ισχυρή εντολή. Η εντολή από, του, του Συμβουλίου από την Κορεπέρ συμφωνήθηκε επίσης στις 13 Ιανουαρίου φέτος και ο τρίλογος ξεκίνησε άμεσα, δηλαδή 1η Φεβρουαρίου. διαπραγματευτική ομάδα συμφώνησε γύρω από ένα πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν να φτάσουμε σε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου. Πολλέ τεχνικέ συνεδριάσει έλαβαν χώρα και προβλέπονται και άλλες έως τις 15 ε, Μαρτίου που είναι και ο τελευταίος τρίλογος. Τρεις λοιπόν τριμερίδες διάλογοι έλαβαν χώρα, ε, σημειώθηκε πρόοδος και σε ό,τι αφορά την πολιτική συζήτηση αλλά και σε ό,τι αφορά το τεχνικό επίπεδο. Πολλά ζητήματα που αφορούν την κινητικότητα των επιχειρήσεων και σχετική οδηγία που επιτρέπουν στι επιχειρήσει να κινούνται διασυνοριακά μέσω ε, συγχωνεύσεων ενώσεων και διαχωρισμών ε, συμφωνήθηκαν ήδη. Ε, το πιο σημαντικό σημείο στην εντολή του Κοινοβουλίου ε, είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του. Δεν θέλουμε να προδικάσουμε βεβαίως τους τελικούς συμβασμούς. Πάντως αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για μια διαδικασία διευκόλυνση των επιχειρήσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις και οι αρχές να έχουμε μια σαφή διαδικασία και απλή ε, για τις συγχωνεύσεις ε, ε, που θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές αναφορές στη διοίκηση, στους εργαζομένους, να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις και δεύτερον ο ρόλος των εξάρτητων εμπειραγνωμόνων σύμφωνα με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν πλέον απλά τον ρόλο του ελεγκτή ε, στο επίπεδο της αρμόδιας αρχής. Οι ψηφιακές πτυχές τώρα, σε ό,τι φορά τη κινητικότητα, ε, θα υπάρξει μια ευθυγράμμιση με τη συμφωνία για την οδηγία σχετικά ε, με τα ψηφιακά εργαλεία. Τώρα, υπάρχει το θέμα του πώς θα αντιμετωπίσουμε τις τεχνητές συμφωνίες και την κατάχρηση αυτών των διαδικασιών από τις επιχειρήσεις αυτό είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί. Ε, δεν μπορεί ο εισηγητή να βρει μια σωστή και αποτελεσματική λύση. Δεύτερον, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εδώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, αποκλίνουν πολύ στις απόψει του. Η ομάδα διαπραγματεύση ε, εξετάζει ένα νέο ξεχωριστό άρθρο για την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων για να εξασφαλίσουμε ότι το παρόν πλαίσιο θα γίνει σεβαστό στα πλαίσια των νέων δικασιών Μετακίνηση μεταφορά επιχειρήσεων. Το θέμα της συμμετοχή των εργαζομένων πάντως παραμένει ανοιχτό. Το Κοινοβούλιο ε, θέλει μια ενισχυμένη προστασία των εργαζομένων και ε, των δικαιωμάτων συμμετοχή του. Η πρόταση της, ε, του Συμβουλίου είναι πολύ πιο κάτω και από την πρόταση της Κομισιόν για την συμμετοχή των εργαζομένων. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια απόκληση. Αυτά από την Evelyn Regner. Βεβαίως μπορώ να τους μεταφέρω κάποια ερωτήματα, αν ε, θέλετε κάτι να ρωτήσετε, κατά λοιπά ε, νομίζω ότι μπορεί να απευθυνθείτε και στο γραφείο τη απευθείας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν φαίνεται να ζητάει κάποιο το λόγο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σημείο 22. Πάλι εδώ αναφορά την προστασία των προσώπων σε ό,τι αφορά την, κατά την παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Η κυρία Ροζιέρ έχει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω τι γίνεται στη διαπραγμάτευση σε ό,τι αφορά την οδηγία για την προστασία των whistleblowers. Avec le, le premier trilogue, le 29 29 ε, Νοεμβρίου ξεκίνησε ο τρίλογο. Είχαμε πολλέ τεχνικέ συναντήσει έκτοτε. Αυτό μα επέτρεψε να φτάσουμε σε κάποιε συμβαστικέ προτάσει. Έγινε μετά ένα δεύτερο τρίλογο την περασμένη εβδομάδα, 14 Φεβρουαρίου, στο Στρασβούργο. Σε γενικέ γραμμέ, ε, το καλό είναι ότι και τα τρία θεσμικά όργανα θέλουν να κλείσουν τη συζήτηση αυτή πριν το τέλο τη θητεία. Καταφέραμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά από σημεία. Ε, την προστασία των τρίτων προσώπων, το θέμα της καλής πίστης, το θέμα της επιλεξιμότητας για την προστασία αυτή. Όμως διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και κάποια σημεία διαφωνίας αρκετά βαθιά που παραμένουν. Και το πιο βασικό είναι το θέμα της ιεράρχησης. Ε, στην πρόσθεση της Κομισιόν προβλέπονται ε, τρεις διάβλοι για τους μάρτυρες μεσαίου συμφέροντος είτε εντό τη επιχείρησης είτε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι δημόσιες αρχές και ε, τρίτος διάβλος ο τύπος. Ε, και εδώ η Κομισιόν στην αρχή της πρόταση πρότεινε να υπάρχει μια, αυστηρή ιεράρχηση των διάβλων, να ξεκινάει πάντα δηλαδή ε, από την ίδια την επιχείρηση, την προσπάθειά του ε, ο Μάτρε δημοσίου συμφέροντος, εδώ το Κοινοβούλιο διαφωνεί κάθετα εμείς έχουμε μια πολύ ισχυρή εντολή, όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ομόφωνα από την ομάδα νομικών υποθέσεων που λέει η εντολή μας ότι στις πιο σοβαρές περιπτώσεις όπου η ίδια η επιχείρηση, την αφορά την την επιχείρηση, όταν το κείμενο το ίδιο θέλει να, να αποφύγουμε ε, να υπάρξουν ε, αντίπεινα για τον άνθρωπο αυτό, το να τον αποχρεώνουμε να περάσει πρώτα από την επιχείρηση είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή τον εκθέτουμε άμεσα σε αντίπεινα. Εδώ η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφέστατη και ευθυγραμμίζεται και με τι συστάσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη, την οποία προσυπέγραψαν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη, που είναι και στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν ε, συνεπεί, θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε αυτέ τι τάσει τι οποίε υπογράψαμε. Να προσθέσω ότι την περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια σαφή έκκληση ε, από 75 ΜΚΟ ευρωπαϊκέ, την Ένωση Δημοσιογράφων, Transparency International, όλοι αυτοί συμμετέχουν στην προστασία των ματήρων δημοσίου συμφέροντο με τον ίδιο άλλο τρόπο και ζήτησαν από το Συμβούλιο να ευθυγραμμιστεί με τη θέση του Κοινοβουλίου. Επίση, από ό,τι ξέρουμε, ατύπω τουλάχιστον, ότι στο Συμβούλιο δεν υπάρχει μία ενιαία θέση. Υπάρχουν τρει θέσει που συνεπάρχουν. Μία σκληρή θέση, την οποία περισπέζει το Συμβούλιο σήμερα, μία μέση θέση, όπου υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη, τουλάχιστον πέντε, που ανταποκρίνεται στη θέση ε, του Κοινοβουλίου και υπάρχει μια ακόμα πιο ευέλικτη θέση ε, που προέρχεται από μια χώρα που βεβαίως που έχει μακρά ε, παράδοση στην προστασία των μαρτύρων του που πάει ακόμα πιο πέρα από αυτά που λέμε εμείς. Εμείς πρέπει να μείνουμε πάντως στην εντολή μας διότι νομίζω είναι και πιο ισορροπημένη και αυτό που προσπαθήσουμε να κάνουμε στη διαπραγμάτευση. Τώρα ένα άλλο σημείο διαφωνίας όπου επίσης υπάρχει μεγάλη απόκληση είναι το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Και εδώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν δύο προσεγγίσεις εντελώ διαφορετικέ. Το Συμβούλιο θέλει να περιορίσει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Σα θυμίζω ότι και στην έκθεση πρωτοβουλία αλλά και στι εργασίε μα θελήσαμε, και αυτό ήταν και το νόημα τη πρόταση τη Κομισιόν, μια οδηγία όσο γίνεται πιο ευρεία, όσο γίνεται πιο οριζόντια για να εξασφαλίσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη προστασία. Το, το Συμβούλιο όμω περιόρισε το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, εμεί την εντολή μα το διαβρύνουμε Και έχουμε προσθέσει δύο ακόμα νομικέ βάσει ε, που αφορά την προστασία του κοινωνικού δικαίου, των συνδικών εργασία, ε, την προστασία δηλαδή, των εργαζομένων. Και καλό είναι εδώ να θυμίσουμε ότι και για το θέμα αυτό είχαμε σκάνδαλα μέσω μαρτύρων δημοσίου συμφέροντο που αποκαλύφθηκαν μέσω αυτών των μαρτύρων για τι συνθήκε εργασία στο McDonald's, στην Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτέλεσαν αντικείμενο ε, βίντεο για τον κίνδυνο στη, για την ακαιρεότητα των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία να την ε, αγνοήσουμε, ενώ δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, ε, δεν υπάρχει λόγος σε να μην προσθεθεί και αυτός ο τομέας αρμοδιότητας στο πεδίο εφαρμογή ε, της προστασίας που παρέχει η οδηγία. Λοιπόν, δύο αυτά, τα δύο λοιπόν ζητήματα που υπάρχει μεγάλη, αντί, μεγάλη αντίφαση, δύο είναι μόνο, αλλά είναι σοβαρά. Ελπίζουμε να κλείσουμε του τριμερεί διαλόγου την πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρουμε. Υπερασπιζόμαστε την βέβαια πάντα με στεναρότητα την εντολή του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, ο κ. Καβαντά έχει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα στους συναδέλφους. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, χωρίς καμία επιφύλαξη και ε, ειλικρινά την κυρία Ροζιέρ για το έργο της, διότι ορισμένε φορές η θέση του Κοινοβουλίου ε, και το πώς ε, λαμβάνεται υπόψη η θέση ε, στον τρίλογο δεν ανταποκρίνεται στις προσωπικές θέσεις της κυρία Ροζιέρ, όμως έδειξε, επέδειξε έτσι ένα πνεύμα συμβασμού και αυτό είναι ευφυές, διότι έτσι μπόρεσε να επιζήσει το έγγραφο αυτό, το κείμενο αυτό. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε, συμφωνώ μαζί σας κυρία Ροζιέρ, ε, θα πρέπει οι θεσμοί, ιδιαίτερα το Συμβούλιο, να μην ε, ε αφαιρέσουν κάθε περιεχόμενο από την πρόθεση του Κοινοβουλίου. Υπάρχει αυτή, η, αυτός ο πειρασμός, αυτή η θέση, η μέση θέση την οποία ακολουθήσαμε όλοι πίσω από εσά, μας επιτρέπει ε, ε να που με το προφανές ε, ότι πρέπει εμείς στην Ευρώπη να προστατεύσουμε ε, τους μάρτυρες μουσείου συμφέροντος οι οποίοι παντού αλλού στον κόσμο βάλλονται από διάφορες ε, ε δυνάμεις πολιτικές, οικονομικές ε, ε στον παρακευτικό τομέα παραδείγματος χάρη μιλάμε για ζητήματα για τα οποία πρέπει να μάθει πρέπει να τα μάθει το ευρύ κοινό για να μπορούν να παίρνουν και αποφάσεις με πιο εμπεριστατωμένα να γνωρίζουν οι πολίτες δηλαδή να παίρνουν αποφάσει του ε, όλα τα στοιχεία. Θα σα υποστηρίξουμε λοιπόν μέχρι τέλου. Ο κύριο Ντυρό, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, λίγα γαλλικά ακόμα για το θέμα αυτό ε, που μα ενδιαφέρει όλους νομίζω ε, δύο λόγια. Ε, να πω πρώτα ότι η Βιρζινή Ροζιέρ, ο Ζωμαρή Καβαντά, αλλά και οι άλλοι βουλευτές είναι εξαιρετικά αλληλέγγυοι στο ζήτημα αυτό και αυτό είναι προς τιμή ε, του Κοινοβουλίου σημαντικός φάκελος. Όλοι έχουμε καταλάβει ε, ότι θα πρέπει ε, να μπορέσουμε να το περάσουμε αυτό πριν τις εκλογές θα είναι ένα ωραίο, ένα ωραίο μήνυμα που θα δώσουμε και κάτι το οποίο, το οποίο λυπάμαι ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια πιστοχώρηση της Κομισιόν πρέπει να το πω αυτό η Κομισιόν έχει επαναχωρήσει που τελικά εδώ, σε αυτή τη φάση των έχει πάρει θέση. Ενώ ο κ. Τίμερμανς άλλα μας είχε πει, αρχικά μας είχε πει ότι θα υποστηρίξει τη θέση του Κοινοβουλίου, τώρα βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεγγίζει το Συμβούλιο και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Το, η Κομισιόν ουσιαστικά εγκαταλείπει τον αμερόληπτο αντικειμενικό ρόλο του, ρόλο του διευκολυντή είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα για, το, για τη Βυζνή Ρωσία και το έργο της και ε, νομίζω ότι όλα θα παιχτούν ε, εκεί στο ζήτημα του κατά πόσο πρέπει να προστατεύεται ο μάτια δημοσίου συμφέροντος ακόμα και όταν έχει πραγματοποιήσει κάποια παράβαση για να μπορέσει να έχει τα αποδεικτικά στοιχεία στη διάθεσή του. Αυτό ήθελα να πω. Είναι σημαντικό. Πρέπει η Κομισιόν να έρθει πιο κοντά στο Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Λεμπρετό, έχει το λόγο. Είναι ένα κείμενο το οποίο από ό,τι φαίνεται έτσι προκαλεί πάθη στους Γάλλους. Εμεί έχουμε βεβαίω στη Γαλλία με νομοθεσία που προστατεύει του μάτι μας όμω δεν είμαστε εγωιστέ. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και αυτή να χαίρει αυτή τη προστασία. Ε, την Ευρώπη των Εθνών θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, δεν θα τσακωθούμε τώρα γι' αυτό. πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ε, έχει φανεί ότι αυτό χρειάζεται. Το κείμενο αυτό είναι καλό σε γενικές γραμμές, συμφωνούμε στα βασικά για την προστασία των παραβάσεων ε, του δικαίου της Ένωσης, δημόσια υγεία, προστασία του καταναλωτή, ξέχλυμα χρήματος. Τώρα, κατά πόσο να πάμε παραπέρα, δεν ξέρω αν πρέπει να αποτελέσει αυτό αντικείμενο διχόνοιας και αυτό να διακυβεύσει τελικά την έγκριση του κειμένου, εδώ είμαι κάπως επιφυλακτικός εγώ. Ε, τώρα επί της διαδικασίας, όντως, εδώ συμφωνούμε, ακόμα και αν είναι καλό να προβλέπετε μια εσωτερική διαδικασία στις μεγάλες επιχειρήσεις, ε, στις διοικήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να μπορεί κάποιος να απευθύνεται απευθείας στο εξωτερικό. Ε, το έχει δείξει αυτό η εμπειρία. Οπότε εδώ δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε. Η ιεραρχία δηλαδή, δεν πρέπει να είναι πολύ αυστηρή ανάμεσα στην εσωτερική, εξωτερική διαδικασία. Ιδάλω υπάρχει ο κίνδυνο να μην επιβεβαιωθεί ο στόχο μα, να προστατεύσουμε δηλαδή το μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο. Τώρα για τι εγγυήσει του κειμένου, η απαγόρευση αντιπίνων, οι κυρώσει αν εφόσον υπάρξουν αντίπεινα, η συνδρομή που πρέπει να δοθεί από τι αρχέ στον ε, μάρτυρα, όλα αυτά πολύ καλά αν είναι κάτι που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, στα πλαίσια μιας ε, ίστατης διαπραγμάτευσης ε, νομίζω ότι θα πρέπει ε, περισσότερο να εμπερασπιστούμε την ιδέα ε, του να μπορεί να υπάρχει μια παρέκκληση στην εσωτερική διαδικασία και όχι να ζητήσουμε ε, πάση θυσία επέκταση του πεδίου εφαρμογή του κειμένου. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Αν δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, να πάρουμε τουλάχιστον τα πιο σημαντικά. Ευχαριστώ κυρία Γιούτελαντ. Πρέπει να μιλήσετε και εσείς γαλλικά τώρα. Όλοι γαλλικά μιλάνε εδώ. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα καταρχάς όπως όλοι ανέφεραν να συγχαρώ την εισηγήτρια ε, κυρία Χωσιέρ για την σημαντική της εργασία καθώς πρόκειται για σημαντική ε, εργασία για τη δημοκρατία, υπέρ της δημοκρατίας. Γνωρίζουμε ότι πολλοί κάνουν σημαντικές θυσίες για τη δημοκρατία, υπέρ της δημοκρατίας γιατί και εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Εμείς έχουμε έναν, έχουμε ένα, μια νομοθεσία ε, που χρονολογείται και 200 χρόνια ε, για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος τους ε, έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν άμεσα στον τύπο προστατεύονται ενάντια σε μέτρα σε αντίπεινα και μπορούμε έτσι να τους προστατεύσουμε. Αυτό είναι ε, τα κατώτατα όρια προστασίας εξάλλου. Μπορούμε, να, αν θέλουμε, να προσθέσουμε. Και γι' αυτό και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι ότι συζητώνται οι, ε, τα μέτρα αυτά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Συχνά πρόκειται για πολύ εθνικές εταιρείε εξάλλου για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην περιορίζονται αυτά που ήδη έχουμε στη δική μου χώρα, όπως όντως έτσι προβλέπετε. Θα ήθελα να τονίσω και τα όσα τονίσατε για την τελική προσέγγιση και την ιεραρχία των αναφορών. Ε, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η διάβλη είναι επαρκής και ότι δεν ζημιώνουν, δεν βλάπτουν ε, και για μας όπου τα συνδικάτα έχουν τόσο σημαντικό ρόλο είναι κάτι που θα θέλαμε να συνεχίσουμε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ειδικά τα ε, συνδικάτα στην αναφορά ε, σφαλμάτων ή σκανδάλων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Ροζιέρ. Εάν δεν υπάρχει άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα, ήθελα να ξαναπάρω το λόγο για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη στήριξή τους. Είναι αλήθεια, ε, όλη η, η ομάδα, των η διαπραγματευτική ήταν εξαιρετικά αλληλεγγύα και ήταν μεγάλη μου ευχαρίστηση να διαπραγματευτούμε από αυτές τις συνθήκες, αν και θα ήθελα περισσότερη κατανόηση από τους άλλους θεσμούς. Αλλά να πω και να επιβεβαιώσω τη σημασία του συνόλου των ε, μαρτύρων ε, δημοσίου συμφέροντος και να θυμίσω ότι στο πλαίσιο του, εδώ ε, μέσα στο Κοινοβούλιο διοργανώνεται μια έκθεση για τα θύματα του μεδιατόρ που είναι ένα σκάνδαλο υγείας, έχει, γίνει, έχει λάβει χώρα στην Γαλλία, θα δεχθούμε τον του μάρτυρε δημοσίου συμφέροντος, καθώ και το, θα ακούσουμε τη μαρτυρία ενός από τα θύματα, γιατί ξεχνάμε συχνά ότι πίσω από αυτές τις καταχρήσει υπάρχουν πάντοτε θύματα και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για θύματα που έχουν νιώσει στο πετσί τους το ότι έχει συμβεί. Είναι μια έκθεση λοιπόν που παρουσιάζει τα πρόσωπα των θυμάτων, ε, και μας επιτρέπει να επιμένουμε ακόμα μια φορά για τον ουσιώδη ρόλο των ε, μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος για υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και υπέρ της λειτουργίας της δημοκρατίας. Την τρίτη την επόμενη 26 το μεσημέρι. Ε, ξεκινάει αυτή η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Άλλος δεν ζητά το λόγο για αυτό το θέμα, οπότε τέλος... ψηφιακή νέα αγορά και πνευματικά δικαιώματα. Το λόγο έχει ο κύριος Βόσα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι την περασμένη Τετάρτη το βράδυ στο Στρασβούργο καταλήξαμε στη συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Βέβαια να πω ότι από τις ε, τέσσερις προγραμματισμένες ώρες συνεδριάσαμε 13. Και πραγματικά θέλω να συγχαρώ εκείνους ε, που άντεξαν και δούλεψαν σκληρά, συναδέλφους, ε, βοηθούς, ιδιαίτερα τη γραμματεία η οποία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για να μας βρει αίθουσα, για να μας εξασφαλίσει η διερμηνία. Γι' αυτό λοιπόν ένα Ιδιαίτερα ευχαριστώ στη Γραμματεία από όλους εμάς που καταφέρατε να μας παρέχετε την δυνατότητα της ε, συνεδρίασης όλη μέρα έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας. Ε, πρώτα, να πω ότι σε γενικές γραμμές τα άρθρα 13 για το κενό αξιών, 11 για την προστασία των δικαιωμάτων, 14, 16α και 3α. Ε, ήταν άρθρα που συζητήθηκαν ε, μαζί. Η, καταλήξαμε σε συμφωνία για όλα αυτά και μετά υπήρξαν βέβαια ορισμένες ε, επιμέρους λεπτομέρειες τις οποίες χρειάστηκε να συζητήσουμε όλη τη μέρα. Ε, η μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αναφέρεται ιδιαίτερα στο άρθρο 13. Εδώ υπάρχουν ορισμένες ε, προϋποθέσεις για την ε, λογοδοσία, για την ευθύνη μιας επιγραμμικής πλατφόρμας. Προσπαθήσαμε αυτό να μπει και στους ορισμούς στο άρθρο 2 παράγραφος 5. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι χρειάζεται να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση. Γι' αυτό λοιπόν να τονίσω ότι δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι πλατφόρμες το άρθρο 13, αλλά μόνο οι πλατφόρμες οι οποίες χρησιμοποιούν έργα με, ε, τα οποία έχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται. Το περιεχόμενο λοιπόν θα αποθηκεύεται και θα προετοιμάζεται καταλήλως έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο στο κοινό. Αυτές οι περιπτώσεις ε, λοιπόν αναφέρονται στο άρθρο 13. Επίσης υπάρχει ένας αρνητικός κατάλογος στο άρθρο 2 παράγραφος 5 για πλατφόρμες ε, όπως εκείνες ε, open source, ε, όπως η Wikipedia για παράδειγμα, οι επιγραμμικές εγκυκλοπαίδειες, στις οποίες οι ίδιοι δημιουργοί ανεβάζουν τα δημιουργήματά τους και δεν συμπεριλαμβάνονται πλατφόρμες όπως το Dropbox, ας πούμε, όπου ο καθένας μπορεί να ανεβάσει περιεχόμενο, το οποίο όμως δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό. Επίσης, συζητήθηκαν όλες ε, οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 14, οι πλατφόρμες για επιγραμμικές γνωριμίες, για παράδειγμα. Συζητήθηκαν με πολλές λεπτομέρειες λοιπόν αυτά τα επιμέρους στοιχεία για να δούμε τι θα κάνουμε έτσι ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται τα πάντα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Επίσης υπάρχουν ορισμένες ε, περιπτώσεις για τις οποίες επέμεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οδηγηθούμε σε συμφωνία και ε, να, προστατεύονται, να προστατεύεται το περιεχόμενο το οποίο ανήκει σε κάποιον ε, δημιουργό που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια του ε, κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων για να ε, δημοσιεύεται το περιεχόμενο αυτό στην εκάστοτε πλατφόρμα. Μετά, στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη έγκριση του δημιουργού, η πλατφόρμα θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να ενημερώνει τον ε, κάτοχο των ε, πνευματικών ε, δικαιωμάτων ή να μην ανεβάζει περιεχόμενο που προστατεύεται. Μετά, έργα τα οποία ήδη έχουν δημοσιευθεί αλλού. Θα πρέπει να απομακρύνονται ε, από τις ε, πλατφόρμες αυτές εφόσον ε, προστατεύονται. Υπάρχει αυτή η κοινοποίηση από αφαίρεσης δηλαδή, notice of removal. Και εδώ να πω ότι αυτό ήδη προβλέπεται στην νομοθεσία. Τώρα, όλες αυτές οι διαδικασίες, αυτά τα βήματα που ανέφερα, εάν οι πλατφόρμες τα τηρήσουν όλα, τότε δεν θα ε, είναι υπόλογες ε, νομικά για το περιεχόμενο. Προσπαθήσαμε λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα τέλος, να ολοκληρώσουμε τις ε, εργασίες μας. Γι' αυτό λοιπόν και συζητήσαμε το ποιος θα έχει την ε, τελική ευθύνη. Μετά, στο άρθρο 13 υπάρχει και μία εξαίρεση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στο 13.4α προβλέπεται επίσης και μία ελάφρυνση και κάποια ελαφρυντικά στοιχεία για, του, για τις πολύ πολύ μικρές πλατφόρμες ε, που αποτελούνται από έναν ε, χρήστη ας πούμε που δεν έχουν μεγάλο κύκλο εργασιών ε, μέχρι 5 εκατομμύρια επισκέψεις μηνιαίως. Και αυτό μέσα σε διάστημα τριών ετών. Οι ευθύνες λοιπόν της πλατφόρμας αυτής θα είναι περιορισμένες θα είναι υποχρεωμένες μόνο να ζητούν ε, μία άδεια από τον δημιουργό και θα αρκεί μία ειδοποίηση του δημιουργού για να αφαιρεθεί το περιεχόμενο από την πλατφόρμα. Εδώ με το Συμβούλιο συγκρουστήκαμε κάπως για ε, τις εξαιρέσεις ε, που αφορούν το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες Ο χρήστης λοιπόν θα πρέπει να προστατεύεται επίσης ε, όταν ε, ανεβάζει περιεχόμενο που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Εδώ αναφερόμαστε στα διάφορα memes, όμως υπάρχουν, υπάρχει περιορισμένη ευθύνη για τις ε, πλατφόρμες. Όταν ας πούμε δημοσιεύονται σατυρικά, σατυρικές εικόνες, αποσπάσματα, διάφορα memes, τότε η, η ευθύνη της ε, πλατφόρμας θα είναι περιορισμένη. Σε γενικές γραμμές λοιπόν αυτά ως προς το άρθρο 13 είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά τελευταία στα μέσα ενημέρωσης και είναι σημαντικό να γίνεται η σωστή παρουσίαση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 11, όπου υπάρχει το ε, δικαίωμα προστασίας για τους ε, εκδοτικούς οίκους. λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Συμβούλιο με, τις, ε, την ισορροπία των δυνάμεων δεν καταφέραμε να ε, περάσουμε τη θέση μας. Ε, επικεντρωθήκαμε στην ιδιωτική χρήση, μη εμπορική χρήση δημοσιευμάτων τύπου. Καταφέραμε να εστιάσουμε στα μικρά αποσπάσματα, very short excerpts, λίγες λέξεις δηλαδή, καταφέραμε να να περάσουν αυτά έτσι ώστε οι δημοσιογράφοι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ήθελε πολύ να επικρατήσει το Συμβούλιο. Θα το, το συστήσαμε όμως τώρα στο 16α. αναφερόμαστε στην ε, επαρκή αποζημίωση. Εδώ να σας πω πως ε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κοντέψαμε να φτάσουμε σε αδιέξοδο ειδικά από την πλευρά του Συμβουλίου. Όμως καταφέραμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους ε, μικρούς εντό εισαγωγικών δημιουργούς να έχουν τη δυνατότητα αποζημίωσης ε, για το έργο τους. Και σε γενικέ γραμμές ε, να βελτιώσουμε τη θέση των ε, καλλιτεχνών και των μεμονωμένων μικρών δημιουργών σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ενημέρωσης, τις της διαφάνειας με σκοπό Α, να σας πω επίσης ότι προβλέπεται και το ενδεχόμενο διαιτησίας ε, σε περίπτωση διαφωνίας, έτσι ώστε ο καλλιτέχνης να ε, λάβει την ε, αποζημίωση που πρέπει. Και εδώ υπήρχαν δύο προβληματικά σημεία, τα οποία έπρεπε να επιλύσουμε. Το ένα αφορούσε τα καταποκοπή ποσά για την αποζημίωση λοιπόν ε, ενός καλλιτέχνη και το άλλο ήταν θέμα διατύπωσης για τους ε, διάφορους μηχανισμούς που υπάρχουν στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να οδηγηθούν οι δύο πλευρές σε ένα συμβασμό. Μετά ε, συζητήθηκε το data mining στο άρθρο 3 και 3α στο άρθρο 3 περιγράφεται αυτό που ήδη γνωρίζουμε και ήδη εφαρμόζεται ότι δηλαδή προβλέπεται μια δυνατότητα data mining ε, για τους ε, επιστήμονες, για τους ερευνητές. Στο 3α αυτό που κάναμε είναι να, αφορεί, να αφορά αυτή η δυνατότητα και το ψηφιακό περιεχόμενο. Βέβαια, εδώ προβλέπονται και κάποιες εξαιρέσεις για την ε, ιδιωτική ή εμπορική χρήση. Εδώ είναι υποχρεωτικό τα κράτη-μέλη να προβλέπουν και αυτήν την ε, δυνατότητα και προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό της ε, ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Και προσπαθήσαμε λοιπόν ε, να προστατεύσουμε το έργο του δημιουργού. Μετά να σας πω επίσης ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο και η ισορροπία των δυνάμεων είναι προβληματική. Υπάρχουν δύσκολες ισορροπίες. Είναι δύσκολο να οδηγηθούμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα Και το είδαμε και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο από πέρυσι το καλοκαίρι ε, που συζητάμε αυτό το θέμα. Η συζήτηση είναι συναισθηματικά φορτισμένη, υπάρχουν διαφωνίες. Νομίζω όμως πως ε, στο τέλος τα καταφέραμε και βρήκαμε αυτές τις ε, λεπτές ισορροπίες και εδώ αλλά και στο Συμβούλιο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο Συμβούλιο. Ελπίζω λοιπόν πώς καταφέραμε να βρούμε αυτές και να κρατήσουμε αυτές τις λεπτές ισορροπίες για την προστασία των ε, δημιουργών. Ελπίζω λοιπόν να κάναμε κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση για να προστατεύσουμε τους ε, κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων, τους ε, δημιουργούς και θεωρώ ότι οι εξελίξεις ε, στην ψηφιακή τεχνολογία απαιτούν και εμείς να κάνουμε το έργο μας, να κάνουμε τα πάντα για να προσαρμοστούμε. Σε γενικές γραμμές βέβαια, να σας πω ότι προσπαθήσαμε να περιγράψουμε πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν, διότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη για ε, διευκρίνηση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία βάση. Αυτά λοιπόν προς το παρόν και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ κυρία Μπρέντα, έχει το ε, λόγο. Πολλοί έχουν στήσει το λόγο, οπότε σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, να μην χρειαστεί να σας κόψω εγώ στις ομιλίες Κυρία Μπρέντα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα την εντύπωση ότι η συνεδρίαση θα κρατήσει μέχρι τις 12.30. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως πρέπει να αφιερώσουμε στο θέμα αυτό το χρόνο που ε, του αρμόζει, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι τελευταία φορά εξάλλου που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Έμαθα χθε μόλι ότι προγραμματίστηκε μια έκτακτη συνεδρίαση την ερχόμενη εβδομάδα έτσι ώστε να ολοκληρωθεί συμφωνία στον τριμερή διάλογο για να, περάσει, για να φύγει το θέμα αυτό από εμάς, όμως δεν έχουμε κάποιο κείμενο. Ε, βέβαια, αυτή η βιασύνη έχω την εντύπωση ότι γίνεται για να καθησυχάσει τις φωνές διαμαρτυρίας που προέρχονται από τους ε, πολίτες. Από τότε που έγινε γνωστό το αποτέλεσμα του τριμερούς ε, διαλόγου, μαζεύτηκαν αυθόρμητα στην κολονία χιλιάδες ε, ανθρώπων για να διαδηλώσουν και οι διαδηλωτέ άνοιγαν σε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Πρόκειτο για πολίτες οι οποίοι απευθύνθηκαν στους ε, βουλευτές. Έτσι, ε, έτσι μας έλεγαν. Όμως στην πραγματικότητα η επικοινωνία αυτή είχε γίνει από διάφορα bots. Η διαμαρτυρία λοιπόν ήταν ε, εμφανέστατη. Η διαδήλωση στην Κολομία έκανε σαφές το τι συμβαίνει και τους κινδύνους που υπάρχουν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία έχει επιτευχθεί μετά από πάρα πολλές δυσκολίες. Την πολέμησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπλόκαρε η συμφωνία, κατηγορήθηκε, κατηγορηθήκαμε για δημιουργία όχλου για βρώμικο πόλεμο εν ώψη ευρωεκλογών. Αυτό που βλέπω βέβαια είναι ότι είναι ικανοποιητικό το ότι υπάρχει αντίδραση από το ευρύ κοινό και ότι οι πολίτες είναι ενήμεροι. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο. Καταρχάς, ο τριμερής διάλογος είχε πολλές εντάσεις και οδηγήθηκε σε στα άκρα. Το κείμενο που ψηφίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο ήταν ε, πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο καταλήξαμε. Τον Ιούλιο, λοιπόν, ψηφίσαμε στην Ολομέλεια για τη διαπραγματευτική εντολή και τον ε, Σεπτέμβριο καταφέραμε με πολύ πολύ μικρή πλειοψηφία ε, να συμφωνήσουμε για το άρθρο 13. Όμως στον τριμερή διάλογο έγιναν αλλιώ τα πράγματα. Οι πολλοί μικρές επιχειρήσεις τέθηκαν εκ νέου ε, υποσυζήτηση και συζητήθηκε το διάστημα των ε, τριών ετών. Μιλάμε τώρα για πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούνται από ένα άτομο. Δεν μπορώ λοιπόν να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψήφισε κάτι τέτοιο. Επίσης, τις ε, διαπραγματεύσεις Προσπαθήσαμε να περάσουμε τη θέση μας, όμως ε, ο εισηγητής ε, δεν ακολούθησε τις συστάσεις μας σε ό,τι αφορά το αυτόματο φιλτράρισμα πληροφοριών. Μετά, ε, το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, user-generated content. Εδώ οι εξαιρέσεις που προβλέπονται αφορούν μόνο πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή σάτυρα, παροδία κτλ. Εντάξει, η σάτυρα και τα διάφορα αποφθέγματα που δημιουργούνται ως ε, memes με σκοπό το γέλιο είναι κάτι το οποίο είναι και προσωπικό θέμα. Δεν, νομίζω πως υπάρχει ε, κάποια αντικειμενικότητα σε θέματα γούστου και ως προς το τι πρέπει να επιτρέπεται και τι όχι έτσι ώστε να καταλήγει σε ένα αυτόματο, αυτόματο φιλτράρισμα ή μπλοκάρισμα μιας, ε, ενός μήμ, ενός περιεχομένου. Τώρα οι πλατφόρμες, οι επιγραμματικές πλατφόρμες γνωριμιών δεν συμπεριλαμβάνονται. Εδώ πρόκειται βέβαια για πλατφόρμες οι οποίες έχουν περιεχόμενο προστατευμένο. Όμως, μια φωτογραφία που ανεβαίνει ας πούμε, σε μια πλατφόρμα γνωριμιών όπως το Tinder ε, πρέπει να ε, προστατεύεται. Πρέπει να προστατεύεται από, την, ε, από περιπτώσεις καταχρήσεων. Βέβαια στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία κλέβουν φωτογραφίες από το Getty Images ή από κάτι τέτοιο, αλλά με άτομα που ανεβάζουν δικές τους φωτογραφίες, που έχουν τραβήξει οι ίδιοι, selfies. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς συνδέεται η προστασία των δικαιωμάτων δημιουργού με αυτές τις περιπτώσεις όταν ο ίδιος ο χρήστης δημιουργεί ένα περιεχόμενο. Τώρα, η εξαίρεση για τη Wikipedia. Είναι πολύ σημαντικό η Wikipedia να μην εφαρμόσει διαλογή στο ανέβασμα περιεχομένου, αυτόματη διαλογή, αυτόματο, αυτόματο φιλτράρισμα, αλλά να προστατεύονται οι χρήστες ε, τόσο όσο και το περιεχόμενο. Δεν νομίζω λοιπόν πως ε, αυτή η συμφωνία θα λύσει όλα τα προβλήματα που έχει η Wikipedia. Ήδη οι προσπάθειες που έχουν γίνει για ρύθμιση του θέματος αυτού στη Γερμανία έχουν αποτύχει. Η προστασία λοιπόν των ε, επιγραμμικών υπηρεσιών ισχύει για όλες ανεξαιρέτως. Και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ε, δημοσιογράφων. Δεν σύμφωνο με αυτό, με αυτό στο οποίο έχουμε καταλήξει, ότι μόνο οι freelance, οι ελεύθεροι επαγγελματίε δημοσιογράφοι θα ε, πρέπει να αποζημιώνονται. Εδώ είχαμε την ε, έντονη αντίδραση και διαφωνία διάφορων ε, δημοσιογραφικών ενώσεων. Βέβαια, αυτές οι προσπάθειες για ρύθμιση των δικαιωμάτων της επαρχής υπηρεσιών δεν έχουν καταλήξει σε κάποια θετικά αποτελέσματα. Το αντίθετο θα έλεγα. Τέλος, τα, οι συμβάσεις ολικής εξαγοράς ε, θα έπρεπε να επιτρέπονται. Και αναφέρομαι στο κεφάλαιο για την επαρκή και δίκαιη αποζημίωση. Νομίζω πως ε, το κείμενο μετά τον τριμερή διάλογο έχει αποδυναμωθεί τόσο πολύ ώστε δεν μπορούν να προστατεύσει τους ε, δημιουργούς όσο θα ήθελε. Αυτό λοιπόν από μένα επαναλαμβάνω ότι το κείμενο είναι πολύ αποδυναμωμένο σε σχέση με το αρχικό. Η κυρία Κάουφμαν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πάρω την αφορμή να πάρω την ευκαιρία μάλλον ε, με την αφορμή της συζήτηση αυτή να κάνω ορισμένε ερωτήσει στον κύριο Φως. Η Γιούλια Ρέντα είπε πολλά με τα οποία συμφωνώ. Βέβαια δεν έχω διαβάσει το κείμενο τόσο προσεκτικά όσο εκείνη, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω τα εξή για το άρθρο 11, όπου προσπαθεί να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των ε, δημοσιογράφων, των ε, δημιουργών και ε, να αποζημιώνονται επαρκώς στο ανέβασμα επιγραμμικού περιεχομένου. Ή επίσης διατύπωση στο άρθρο 11 για τη δυνατότητα που έχουν οι εκδότες, οι δημοσιογράφοι και οι δημιουργοί να ε, αποκλείουν την δημοσίευση του έργου τους ε, από ορισμένα από ορισμένες πλατφόρμες. Μετά, άρθρο 11. η ιδιωτική ή μη εμπορική χρήση δημοσιευμάτων από μεμονωμένα άτομα. Η προστασία λοιπόν εδώ έχει εξαιρέσει. Ε, ρωτώ λοιπόν, ο ένας απλός χρήστης του ίντερνετ, τι θα απογίνει όταν τεθεί σε ισχύ αυτή η νομοθεσία. Για παράδειγμα, αν πάρει ας πούμε, ένα απόσπασμα από ένα άρθρο και το μοιραστεί στο ίντερνετ, τι, τι θα απογίνει λοιπόν αυτός ο χρήστης, ο οποίος αναδημοσιεύει ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που διάβασε. Άρθρο 13 τώρα. Ο Άξελ βό ανέφερε ήδη κάποιες εξαιρέσεις για τις επιχειρήσεις, στις οποίες καταλήξαμε, για επιχειρήσεις οι οποίες είναι νεότερες, είναι, είναι, υπάρχουν λιγότερο από τρία έτη, πολύ μικρές, νεοφυείς. Αυτές οι εξαιρέσεις πώς προέκυψαν. Με βάση ποια στοιχεία. Επίσης, έχουμε στοιχεία σχετικά με το πόσες ε, νεοφυείς επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό. Μετά, πάλι για το άρθρο 13, το είπε και η κυρία Ρέντα, αυτά τα τσιτάτα, οι καρικατούρες, η σάτυρα, παροδία, τι γίνεται εκεί. Στο 13.5 αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα εξασφαλίζεται το δικαίωμα στην κριτική, στη σάτυρα, στην ε, παροδία, στην καρικατούρα κτλ. Ερωτώ λοιπόν, πώς μπορούμε με ευρωπαϊκή ρύθμιση να υποχρεώσουμε τα κρατημέλη να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο. Πείτε μου δηλαδή πώς ε, το σκέφτεστε αυτό. Διότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές από κράτος σε κράτος Και αυτός ο κατακαιρματισμός ε, νομίζω πως ε, δεν θα λάβει τέλος, το είδαμε και με την ε, οδηγία της, που ανέλαβε η κυρία Ρέγνερ. Ο κύριος Βόλκιν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά το τέλος του σε διαλόγου ζούμε ένα φαινόμενο άνευ μία τόσο ζωντανή συζήτηση στην οποία συμμετέχουν κυρίως οι νέοι Ευρωπαίοι. Είδαμε ότι κατέβηκαν 2.000 άτομα στο δρόμο στην κολονία για να διαδηλώσουν κατά της ε, νομοθεσίας αυτής. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τους νέους να ενδιαφέρονται για την πολιτική. Αυτό βέβαια που είναι πολύ απογοητευτικό, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο κατηγορούν ορισμένοι συνάδελφοι ότι οι υπογραφές αυτές μαζεύτηκαν από bots και όχι από ανθρώπους. Χειραγωγείται λοιπόν, χειραγωγούνται οι πολίτες. Κατηγορούνται πως ε, η γνώμη τους ε, δεν υπάρχει, πως όλα είναι αέρας. Θεωρώ κυρίες και κύριοι ότι εδώ πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτοί που έχουν κατέβει και διαδηλώνουν δεν είναι όχλος, όπως λέει η Κομισιόν, αλλά οργισμένοι, αγανακτισμένοι πολίτες, οι οποίοι νιώθουν ότι απειλείται ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής τους, της κουλτούρας τους, απειλείται ε, να εξαφανιστεί. Το κείμενο, το οποίο βέβαια να το πούμε και αυτό, δεν έχουμε δει, δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα, έχει πολλά δύσκολα σημεία. Υπάρχει η γενικότερη ανησυχία ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε πλατφόρμες ε, όπως το YouTube, το Twitter, το Instagram, ε, θα αλλάξουν ριζικά. Αυτές οι πλατφόρμες είναι αναγκαίες στην σημερινή κοινωνία της πληροφορίας και νομίζω πως θα είναι τραγικό λάθος να γνωρίσουμε αυτό το γεγονός. Μπορούμε να προσπαθήσουμε βέβαια να αλλάξουμε την πραγματικότητα, όμως αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε κάνει τραγικό λάθος, θα έχουμε χτυπήσει ε, την ε, καρδιά της κουλτούρας ε, των νέων πολιτών. Βέβαια, σίγουρα οποιαδήποτε πλατφόρμα έχει καταφέρει να έχει και εξαιρέσει. Αλλά μιλώ για τις μεγάλες. Αυτές που δεν έχουν εξαιρέσει είναι αυτές που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, αυτές που δεν υπάρχουν. Εδώ υπάρχει αυτή η εξαίρεση για τις ε, νεοφυείς επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με λιγότερο από τρία χρόνια. Τι γίνεται όμως όταν μια τέτοια μικρή επιχείρηση εξαγοράζεται από έναν ε, πολυεθνικό κολοσσό. Εδώ πώς θα αντιδράσετε. Μας λέτε ότι χειραγωγούνται οι νέοι από την Google όμως οι νέοι λένε κάτι άλλο. Λένε ότι η ελευθερία αυτή είναι δική μας και δεν θέλουμε λογοκρισία. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως εδώ δεν ε, πρέπει να μιλάμε για χειραγωγημένο όχλο, αλλά για προσπάθεια θύμωσης. και αυτό να γίνει σαφές. Στο άρθρο 11 φοβάμαι ότι σοβαρές εφημερίδες, σοβαρά μέσα θα προσπαθήσουν να πουλήσουν, ε, να αγοράσουν μάλλον άδειες έτσι ώστε να εξαφανίσουν τους, ε, τα μικρότερα μέσα ενημέρωσης ε, και αυτός που θα αποφεληθεί στο τέλος φοβάμαι πως θα είναι οι ψευδείς ειδήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ έχουμε αντιδράσει με υπερβολή και αυτό είναι αντίθετο στους σκοπούς της οδηγίας. Τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέπετε μια πραγματική εξαίρεση για το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι ίδιοι οι δημιουργοί. Αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο. Όταν αναφέρουμε ότι υπάρχουν εξαιρέσεις θα πρέπει να αναφέρεται επίσης και πώς θα διασφαλίσουμε την ε, διατήρηση των εξαιρέσεων αυτών και την διαπίστωση ότι πρόκειται περί εξαίρεσης. Αυτό το φίλτρο είναι ο φόβος και ο τρόμος. Και μας λέτε ότι δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το φιλτράρισμα στο μέλλον, το αυτόματο φιλτράρισμα και νομίζω ότι εδώ βρίσκεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Σόνα. Thank you, Chair. On the... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το θέμα των bots έχω αποδείξεις ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που μου έστελαν εμένα mail στη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν Σουηδοί και μπορώ να το αποδείξω διότι στο standard email απάντηση είχα ένα βίντεο YouTube που απαντούσε για το άρθρο 11 και το άρθρο 13. Και άρα ένα κομμάτι από αυτούς είδαν το βίντεο και έχω και στατιστικές. Όμως ε, παρατηρήσαμε ένα μικρό πρόβλημα. Υπήρχε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό τουρνουά πρωτάθλημα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Νομίζω πως ήταν το ευρωπαϊκό ή ήταν το παγκόσμιο. Α, ήταν το παγκόσμιο κύπελο. Μπάς περιπτώσει, εγώ που δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο, ήταν ε, το ευρωπαϊκό, το, το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Όταν έπαιζε λοιπόν η Σουηδία ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, Τα ποσοστά στο βίντεο του YouTube, το δικό μου, έπεσαν κατά 60%. Είμαι αρκετά βέβαιος ότι τα bots δεν σταματά να διαβάζουν τα mail τους επειδή παίζει η Σουηδία ποδόσφαιρο στην τηλεόραση. Αλλά οι Σουηδοί το κάνουν. Και βεβαίως Είδαμε και ανθρώπου που δηλώνουν δυο mail, υπήρχαν επικαλύψει, ναι, εντάξει, αλλά βασικά πρόκειται για πραγματική ανησυχία των πολιτών, όπου πολλοί κόσμος έρχεται σε επαφή με τους πολιτικούς, γιατί ενδιαφέρονται για το θέμα και το μελετούν. Οπότε παρακαλώ λάβετε σοβαρά υπόψη τον κόσμο. Επίση, θεωρώ πω είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονό ότι αυτή η πρόταση μπορεί να περάσει γιατί θα βλάψει σοβαρά το ίντερνετ όπω το ξέρουμε μέχρι σήμερα και επίση υπάρχει μέγα κίνδυνο ότι θα βλάψει και την οικονομία γιατί θα κάνει τη ζωή δύσκολη για τις εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του ίντερνετ ώστε να παίρνουν σχόλια, να μοιράζονται πράγματα. Εταιρείες όπως το ε, TripAdvisor και όλοι οι ανταγωνιστές του οι εταιρείε που έχουν φόρουμ ε, με διαφημίσεις, ε, σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις ε, σελίδες τους για να κερδίσουν κίνηση. Πολλοί κόσμος λοιπόν θα επηρεαστεί και πολλοί κόσμος θα θυμώσει όταν θα ανακαλύψει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση τους εμποδίζει να έχουν τι επαφές, να ανεβάζουν πράγματα. Κάποιες φορές είναι παράνομο το να ανεβάσεις περιεχόμενο, αλλά υπάρχει και ο, ένας κακός νόμος ο οποίος τους εμποδίζει. Εγώ είμαι πιο ευρωσκεπτικιστής από ότι πολλοί εδώ. Είμαστε ένας ρεαλιστής, σκανδιναβός, κεντροαριστερός, ε, ευρωπαίος, πολύ μυστήριος για τους ε, Βρετανούς ε, συναδέλφους. Δεν θα τους σχολιάσω αλλά ε, ε, βασικά δεν είμαι ικανοποιημένο με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φω για τη σκληρή του δουλειά και γιατί δείχνει στον κόσμο και στους νέους τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημοκρατικά δυσλειτουργική, υπεροπτική και ε, μπορεί να επηρεάζεται από ε, παλαιωμένες ε, ιδέες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροζιέρα. Εγώ πραγματικά με, με έχει ζαλίσει, με έχει ανακατέψει το ότι ακούω τέτοιες ε, απόψεις εδώ. Έχουμε ακούσει διάφορα λόμπι κάλυψης ε, των μαζών και ε, από, τε, από τις ιδιωτικές εταιρείες. Το λόμπι ή πουλά και καλυμμένα ε, λειτουργεί τους εδώ και μήνες. Οι, τα, οι ομάδες πίεσης είναι η γκάφα. Δεν είναι περάξενο. Φτάνει να δει κανείς σε ποιον ωφελούν τα εγκλήματα. Με ένα κομμάτι της κοινή γνώμης έχει τελικά κινητοποιηθεί ενώ έχει έχει βομβαρδιστεί με μηνύματα προκατηλημένα για μήνες και μήνες. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον, δηλαδή να είναι κανείς τελείως ε, άσχετος με την ε, ψηφιακή επιρροή. Δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες ε, οι οποίοι υπόκειται την ψηφιακή παρέμβαση, αλλά και το επάγγελμα ενός καλλιτέχνη είναι να δημιουργεί. Δεν είναι να σκέφτεται πώς θα διαδοθεί ψηφιακά το έργο του. Άλλοι το σκέφτονται αυτό. Μόνο το πρόβλημα είναι ότι το μόνο που σκέφτονται εκείνοι είναι ε, ε, το δικό του κέρδος, το value gap, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί. Εδώ και χρόνια διαπιστώνουμε ότι η διάδοση των ε, πολιτιστικών έργων και των δημιουργημάτων γίνεται προς όφελος κάποιων μόνο από τον ενδιάμεσον και δεν ωφελούν, δεν, δεν ωφελούν τους δημιουργούς τους. Ακριβώς η ευρωπαϊκή κουλτούρα υποφέρει από αυτό, η οικονομία του πολιτισμού βεβαίως, αλλά και η, η δημιουργικότητα, γιατί οι καλλιτέχνες στερούνται των νόμιμων εσόδων από τα έργα τους και περιμένω να δω ποιες είναι οι συμβιβαστικέ λύσεις που έχουν επιτευχθεί στη διάρκεια του τριμερούς. Ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες υπήρχε μεγάλο αίτημα, δηλαδή το άρθρο 14 που θέτει το θέμα της αμοιβή των καλλιτεχνών, να δούμε αν αυτό υπάρχει στις συμβαστικές. Αυτό ήταν ένα έντονο αίτημα της ομάδας μας, αλλά πρέπει να δούμε το κείμενο με τις λεπτομέρειές του. Ε, εν πάση περιπτώσει, εάν είναι στον τελικό συμβιβασμό, θα είναι μια νίκη γιατί, και θα είμαι πολύ ικανοποιημένη, γιατί αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί είναι οι καλλιτέχνες και οι πολίτες δηλαδή. Εάν οι δημιουργοί δεν μπορούν πια να δημιουργήσουν, μπορεί να τους δώσουμε όσου ενδιάμεσου ψηφιακού θέλουν, αλλά δεν θα φτιάχνουν πια έργα. Ε, αυτά όσον αφορά το περιεχόμενο και την εργασία, τη δέσμευση που θα πρέπει να έχουμε για την ευρωπαϊκή μας κουλτούρα και τους ευρωπαίους καλλιτέχνες. Γιατί εγώ προτιμώ να στηρίξω τους Ευρωπαίους ε, ε, καλλιτέχνες από ότι τους ε, ψηφιακούς γίγαντες, τους Αμερικανούς, οι οποίοι έχουν πραγματικά χαλάσει τη συζήτηση εδώ και μήνες με ψευδείς εκστρατείες, παρεμβαίνουν think tank που χρηματοδοτούν δίθεν τις εκστρατείες, ποιοι βρίσκονται από πίσω, το CCIA, δηλαδή τα αμερικανικά λόμπι που καλύπτουν, ε, συγκαλύπτουν και ε, δείχνουν ότι δήθεν είναι αυθόρμητες εκστρατείες, οι εκστρατείες lobbying, πίεσης. Αυτοί όλοι είναι γραμμένοι και στον, ε, στον κατάλογο του Κοινοβουλίου για τα λόμπι, αλλά βρίσκουν πάντοτε έναν αχυράνθρωπο ή αχυροεταιρεία για να καλυφθούν. Και μπροστά και μπροστά στο Κοινοβούλιο, όταν γινόταν η πρώτη ψηφοφορία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, είχε ένα τεράστιο πανό που έλεγε ότι ε, το ίντερνετ δολοφονήθηκε. Όταν κανείς ακούει, ακούει ξανά και ξανά ότι το ίντερνετ δολοφονήθηκε, ε, όλοι οι που ασχολούνται με το, με, το ίντερνετ λέγανε ότι πάλι θα κλείσουν το RG5 GDP, το GDPR ε, όμως τέθηκε επίσης εφαρμογή και συνεχίζουν να δουλεύουν λέγανε ότι πάει, τελείωσε, δεν θα μείνουν χωρίς δουλειά. Αυτά τα μηχανήματα είναι στη ΣΥΠΑ. Όταν βλέπουμε τα, Twitter, τα tweet που στέλνονται όλο το καλοκαίρι. Ναι, ορισμένα έρχονται ίσως από τη Σουηδία. Αλλά όταν βλέπουμε τις στατιστικές, 71.000 tweet που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 80.000 από τη Washington. Πολλοί Ευρωπαίοι, δηλαδή τι είχαν πάει διακοπές στη Washington εκείνη τη φάση. Από το φθινόπερο έχουμε το YouTube που διαδίδει ψευδείς ειδήσει σε όλους τους YouTuber για να τους κάνει να πιστέψουν ότι αυτό που θα ψηφίσουμε θα τους εμποδίζει αύριο μεθαύριο να φτιάχνουν τα βιντεάκια τους. Είναι ψέμα και είναι και σοβαρό γιατί οι συνάδελφοι μίλησαν για τη δυνατότητα της νεολαίας να πολιτικοποιηθεί και να κινητοποιηθεί. Όμως ένας ε, ε, γίγαντας ε, ψηφιακός σαν το YouTube να χρησιμοποιεί τους νέους και να τους χειραγωγεί και να τους πλημμυρίζει με ψέματα είναι πραγματικά απέσιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό όσον αφορά τη δημοκρατική συζήτηση. Προδίδει στην ουσία τους νέους και όχι τους υποστηρίζει. Πιστεύω πως το εύρος, η βία των εξτατιών που ε, ήμασταν εμείς αντικείμενο τους και είδαμε να αναπτύσσονται δείχνουν πως είναι στον καλό δρόμο γιατί η γκάφα φοβούνται και ίσως επιτέλους να επιβάλλουμε την ε, προτεραιότητα της δημιουργίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στους ε, Αμερικανούς γίγαντες. Ευχαριστώ, κυρία Χάουταλα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ βεβαίως είμαι cool Σκανδιναβή. Είμαι φιλοευρωπαία απολύτως και θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για το ότι υπάρχει τόσο μεγάλος διχασμός στο Κοινοβούλιο και στην κοινή γνώμη για αυτή την υπόθεση. Εγώ είμαι πεπισμένη πως θα ήταν πολύ καλό οι συγητέ και οι σκιώδεις συγητέ να ακολουθήσουν τους νέους, το νέο κανονισμό και να δημοσιεύσουν με ποιους συνομιλήσαν στη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, γιατί τώρα φτάνουμε στο τέλος. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι, αρκεί κανείς να προσαρτήσει ένα δελτίο στην έκθεση, αφού περιμένουμε την υποδομή online να φτιαχτεί. Αυτό που σημαίνει είναι ότι γίνεται αυτή η συζήτηση σε μια ε, μισοάδια αίθουσα ενώ πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα αυτής της θετίας που σύντομα τελειώνει. Η συζήτηση αυτή δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, γιατί δεν έχουμε το κείμενο για να συζητήσουμε. Και αυτό που άκουσα εγώ από τη ε, μέσα είναι ότι υπάρχουν κάτι ασαφείς και σκοτεινοί ορισμοί και διατυπώσεις. Φοβούμε λοιπόν ότι το δικοστήριο θα έχει πολλή δουλειά για να ε, δώσει τη σωστή ερμηνεία, ας πούμε, στο πώς μπορεί ε, να βελτιώσει μάλλον η πλατφόρμα να αποδείξει ότι έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να αφαιρέσει το προστατευόμενο υλικό και τι σημαίνει πολύ σύντομο κείμενο. Οι νομοθέτες δεν χρησιμοποιούν κανονικά τέτοιες εκφράσεις, γιατί μετά μόνο το δικαστήριο μπορεί να εξηγήσει τι σημαίνει κάτι τέτοιο και αυτό είναι πολύ ατυχές. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν από τη Γιούλια Ρέντ και τον Μαξ Άντερσον, καθώς και η εξαίρεση των νεοφιών επιχειρήσεων από την υποχρέωση είναι χωρίς νόημα, διότι Πολύ λίγοι μπορούν να ξεφύγουν από αυτά τα κριτήρια, δηλαδή κύκλος εργασιών λιγότερο από 10 εκατομμύρια ετησίω, λιγότερο από 5 εκατομμύρια μηνιαίοι επισκέπτες στο δίκτυο και ε, ήταν σωστό ότι ένας από τους συναδέλφους ρώτησε πόσες ε, νεοφύης startups ξεφεύγουν από αυτές τις υποχρεώσεις. Ε, και όπως είπα, Εμένα με προσβάλλει βαθιά αυτή η προπαγάνδα που δημοσίευσε η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκε σε αυτή η Γιούλια Ρέντα και προσπάθησε να προτείνει να δείξει ότι όλες αυτές οι τη είναι καταπληκτικά για όλα τα μέρη και ότι κάποιοι αλητήριοι προσπαθούν να διαταράξουν αυτή την εργασία. Ε, δεν ήταν εντυπωσιακό που η Κομισιόν χρειάστηκε να αποσύρει αυτό το άρθρο με πολύ αδέξιες εξηγήσεις ότι δεν ήταν πρόβλημα το ότι περιείχε το άρθρο, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι θα μπορούσε κανείς να παρεξηγήσει τα όσα έλεγε και ότι δεν αντικατόπτυζε την γνώμη της Επιτροπής. Αυτό δεν θα πρέπει ποτέ ξανά να συμβεί. Ελπίζω λοιπόν πως θα προσεχθεί πολύ αυτή η υπόθεση στο εμπορία για την Ολομέλεια. Και φυσικά η επόμενη εβδομάδα θα είναι αποφασιστική σημασία για την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Κύριο Ζβιεύκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άλλο ένα επεισόδιο στη συζήτηση αυτή. Ένα σημαντικό ζήτημα, βέβαια, Ήθελα να πω κάποια πράγματα όμως ε, μετά από αυτό που είπε η κυρία Ροζιέρ θα είμαι πιο σύντομος διότι συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε κυρία μου. Σε ό,τι αφορά τώρα τους προηγούμενους ομιλητές αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έγινε έτσι μια προσπάθεια ε, να δημιουργηθεί μια ένταση και όντως είναι ένα θέμα που ε, οξύνει τα πάθη λάβαμε ε, ε, μια έρευνα το καλοκαίρι τα πρόσφατα μιας έρευνας ε, που δείχνει ότι αμερικανικά χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για να προωθηθούν συγκεκριμένοι σκοποί στην Ευρώπη θα μπορούσαμε ποτέ να είχαμε εμεί τέτοιον αντίκτυπο ε, στους Αμερικανούς, στην Αμερικανική κυβέρνηση, να έχουμε λόγο για το τι γίνεται στην Αμερικανική αγορά, είναι απίστευτο. Με τη σειρά όμω. Η κυρία Ρέντα είπε ότι υπήρξε υποστήριξη για τη δεσμευτική εντολή οριακή. 438 υπέρ 246 κατά. Σας φαίνεται πραγματικά οριακή αυτή η διαφορά. Να είμαστε σοβαροί. Άλλη μια προσπάθεια χειραγώγησης θα έλεγα. Χαίρομαι βεβαίως που νέοι άνθρωποι συμμετέχουν ε, σε αυτή τη διαδικασία που ερισπέζεται όχι βέβαια ακριβώς τα συμφέροντά τους προσπαθούμε να υπερασπιστούμε μέρος του πολιτισμού μας. Ε, το ίντερνετ είναι μέρος του πολιτισμού μας. Όχι μόνο των νέων, αλλά και της δικής μου γενιάς. Πώς όμως ε, εμείς ε, οθούμε τους νέους να πάρουν την απόφασή τους. Δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο των εγγράφων των κειμένων. Δεν γνωρίζουν πώς προχωράει η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Μαθαίνουν από εδώ και από εκεί κάποια ε, πληροφοριών. Εγώ θυμάμαι πώς χρησιμοποιούταν η προπαγάνδα στη χώρα μου. Οι νέοι άνθρωποι στη δική μου χώρα διαμορφωνόταν ε, για να χειραγωγούνταν για να μπορούσαν να κατέβουν στον δρόμο και να κάνουν κάτι. Λοιπόν, βλέπουμε τι κάνουν οι Αμερικανικοί τεχνολογικοί γίγαντες, προσπαθούν να, ε, να επηρεάσουν τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου πριν την ψηφοφορία. Τώρα, η λέξη bot, εμένα δεν μου αρέσει και τόσο αυτή η λέξη. Εγώ θα μιλούσα για αυτοματοποιημένη αποστολή συγκεκριμένων μηνυμάτων τα πολωνικά μέλη του Κοινοβουλίου έλαβαν δύο μηνύματα. Δύο. Αυτά τα δύο κείμενα ήταν ολόιδια. Πώς γίνεται αυτό. Τώρα η Τζούλια και εγώ πήγαμε στη Silicon Valley ε, στις ΗΠΑ και να μιλήσουμε για τη start-up. Start-up, δηλαδή μικρές ε, εταιρείες ε, στην αρχική φάση ανάπτυξής τους που χρειάζονται και βοήθεια. Πόσο, για πόσο καιρό όμως είναι μια εταιρεία είναι startup. Ένα χρόνο. Οι Αμερικανοί μας είπαν ότι πέρα από ένα χρόνο αυτές οι εταιρείε είτε αναπτύσσονται περαιτέρω και πλέον επιτυχείς εταιρείε, είτε καταραίουν. Μετά από τρία χρόνια λοιπόν είναι μια απλή μικρομεσαία εταιρεία αυτή. Τρία χρόνια αρκούν. Σαφώς. Τώρα η Τζούλια Ρέντα λέει ότι στις διαπραγματεύσεις ο εισηγητής ε, δεν ασχολήθηκε παρκώς με την ε, διεύρυνση του πεδίου των ε, προθεσμιών για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών. Νομίζω ότι στο έργο μας αυτό που μας, πρέπει να μας απασχολεί είναι το συμφέροντα του χρήστη, του τελικού χρήστη. Πρέπει ταυτόχρονα να υπερασπιστούμε βέβαια στον πολιτισμό μας, να υποστηρίξουμε τις εταιρείε που λειτουργούν σωστά. Οπότε μην πείτε ότι, μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ότι κάποιο δεν θα μπορεί να γράψει ε, μια έκθεση για ένα προϊόν ε, Εγώ μπορώ να δημοσιεύσω ό,τι θέλω και όπως θέλω. Κανείς δεν θα με σταματήσει. Σε κανένα άλλο έγγραφο ευρωπαϊκό δεν έχει περιγραφεί τόσο καλά ο τελικός χρήστης. Όλα αυτά είναι σαφέστατα. Στο άρθρο 13 ε, όταν είναι η διαπραγμάτευση ε, της εντολής. Το άρθρο ήταν ε, μία σελίδα, τώρα είναι τέσσερις σελίδες. Γιατί, γιατί έχουμε καλύτερες, καλύτερους ορισμούς, καλύτερες περιγραφές. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, τα κράτη-μέλη ε, έκαναν μια σελιδα τωρα ειναι τεσσερις σελιδες γιατι γιατι εχουμε καλύτερου ορισμού, καλύτερε περιγραφέ. περιγραφες κατα τη διαρκεια της τα κρατη μελη εκαναν μια προσπαθεια για να εξασφαλίσουν διαφάνεια, σαφήνεια στους κανόνες αυτούς. Βεβαίως συμφωνώ ότι προφανώς ε, δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα πάντα. Δεν μπορούμε να προλέψουμε τα πάντα. Ποιος μπορεί να προλέψει τα πάντα. Ποιος νομικός μπορεί να το κάνει αυτό. Κάποιοι συνάδελφοι λένε ότι πρέπει να το στείλουμε στα, στα σκουπίδια το έγγραφο αυτό, διότι δεν μπορεί να προλέψει, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια. Ακούστε, θα πρέπει να εγκριθεί το έγγραφο αυτό και έτσι θα αποδείξουμε ότι μας ενδιαφέρουν τελικοί χρήστες ε, ή ε, δημιουργοί, οι καλλιτέχνες, η ταυτότητά μας. Δεν πρέπει λοιπόν αυτοί που έχουν τα πολλά τα χρήματα και θέλουν να βγάλουν ακόμα περισσότερα από εμά να μας υπαγορεύσουν το τι θα συμβεί. Ευχαριστώ κύριε Λεμπρετό, έχει τώρα το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, είχαμε εδώ μια τιτάνια ε, μάχη μεταξύ των δημιουργών των Ευρωπαίων που θέλουν ε, εντελώς θεμητά να αμείβονται για τη δουλειά τους και βέβαια από την άλλη έχουμε τις γκάφα που θεωρούν ότι αν ψηφίσουμε αυτό το κείμενο το ίντερνετ θα εκλείψει. Εγώ δεν πιστεύω κάτι τέτοιο βέβαια. Και βεβαίω εγώ υπερασπίζομαι την ευρωπαϊκή κουλτούρα κατά των ορέξεων των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων. Να υπογραμμίσουμε ότι αυτέ οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι μόνο αμερικανικέ, αλλά όλο και πιο συχνά κινέζικέ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ε, επεκτείνονται γκάφα και εκεί. Θα πρέπει λοιπόν εμεί να υπερασπιστούμε την ευρωπαϊκή μα, τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό και την κουλτούρα απέναντι στου Αμερικανού αλλά και του Κινέζου ο τρίλογος από αυτή την άποψη, ο τριμερής διάλογος θα οδηγήσει πιστεύω σε ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί πρόοδο διότι βεβαίως μπορεί να έχουμε επιφυλάξει για το ένα ή το άλλο αλλά είναι προφανές ότι οι δημιουργοί θα προστατεύονται καλύτερα μετά την έγκριση του κειμένου αυτού από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε αυτό είναι πρόοδος. Τώρα για το τεχνικό κομμάτι προφανώς δεν θα είναι όλα τέλεια ακούγοντας τον κύριο Βος ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί. Ε, δεν θα είναι τελείο αποτέλεσμα. Το καταλαβαίνουμε. Έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό το καθεστώ παρέκκληση ότι αφορά τη startup λιγότερο από τρία έτη καλό είναι. Τρία χρόνια είναι παρκή νομίζω για να αναπτυχθούν αυτέ οι εταιρείε. Κατά τα λοιπά, ακούστε, εάν κάποιε διατάξει είναι ασαφείς, ε, το δικαστήριο θα φροντίσει να τα διευκρινίσει αυτά είναι ένα νέο κείμενο το οποίο δεν το γνωρίζουμε κιόλα ακριβώ. θα πρέπει να το δούμε όμως ως ένα πρώτο βήμα αποφασιστικό βήμα αλλά θα υπάρξουν και άλλα θα ερμηνεύσει όλα αυτά και το δικαστήριο και στη συνέχεια με βάση τις ατέλειες που θα εντοπιστούν θα έχουμε κάποιο νέο κείμενο αυτό θα το κάνουν βέβαια άλλοι όχι εμείς ε, εγώ πάντως χαίρομαι που συμμετείχα σε αυτή τη μάχη ε, για την ευρωπαϊκή κουλτούρα, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό κατά και αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ τον κύριο Λεμπρετό. Η κυρία Ρέντα θέλει να επανέλθει. Παρακαλώ, σύντομα όμω. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα ζητούσα το λόγο αν δεν με προκαλούσε ο κύριος Σβιέφκα αναφέροντας ε, λόγια όπως χειραγώγηση και ψέματα. Να σας ε, βάλω τα πράγματα λοιπόν στη σωστή σειρά. Είπα ότι η πλειοψηφία ήταν ε, στενή το Σεπτέμβριο. Είπα 366 ψήφοι υπέρ, 297 κατά. Πάνω από 70 ψήφοι ήταν ε, αποφάσιστον των. Αυτό λοιπόν για μένα καθιστά μια ε, στενή ε, πλειοψηφία. Κανείς δεν μίλησε για χειραγώγηση. Και φυσικά Πολλοί ευρωβουλευτέ στο τέλο ψήφισαν υπέρ τη έναρξη ε, διαπραγματεύσεων, όμω κύριος... Ε, όμως πιστεύαμε ότι ο κύριο Φω θα λάβει σοβαρά υπόψη την κριτική που είχε ασκηθεί και θα προσπαθούσε να ε, τροποποιήσει το κείμενο. Όμω αποδυναμώθηκε πάρα πολύ, ιδιαίτερα ει βάρο των μικρών επιχειρήσεων. Για μένα το θέμα δεν είναι οι startups, οι νεοφύης επιχειρήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλέ πολύ μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε θα υποφέρουν με την έγκριση ενό τέτοιου κειμένου. Υπάρχουν πλατφόρμες ε, που ε, τις χειρίζεται ένα ένας χομπίστας ο οποίο το κάνει από προσωπικό ε, μεράκι. Όταν λοιπόν αυτή η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται ένα, θα κατηγορηθεί για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία, θα καταστραφεί, θα κλείσει. Το ίντερνετ δεν θα πρέπει να αποτελείται μόνο από ε, κολοσσούς ε, και ε, startups, ε, επιχειρήσεις. Δεν είπα επίσης ότι στο ε, μέλλον, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δεν θα μπορεί ο καθένας μας να γράψει την άποψή του, δεν θα μπορεί να ανεβάσει, δεν θα να μιλήσει. Αυτό που είπα είναι ότι τα αυτόματα φίλτρα που θα αποφασίζουν δεν θα είναι σε θέση να κρίνουν πότε ένα περιεχόμενο είναι, ε, παραβιάζει τους ε, κανόνε και πότε όχι και θα μπλοκάρουν αυτόματα ενδεχομένως τα λάθο πράγματα. Επίση, για το streaming όταν ε, πρόκειται για, μια, για ζωντανή αναμετάδοση ενός παιχνιδιού, δεν θα έχει τη δυνατότητα κάποιος ε, να σχολιάζει ζωντανά την ώρα που γίνεται, αλλά μετά από 24 ώρες. Κατόπιν εορτής δηλαδή, ποιο νόημα θα έχει. Τώρα, η κυρία Χάουταλα έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είπε ότι πρέπει να ε, δούμε ακριβώς τι γίνεται με τα λόμπι και ποιος επηρεάζεται. Και γι' αυτό λοιπόν ζήτησα να δημοσιευτεί ο κατάλογος ε, των ε, λόμπι. Το ζήτησαν και πολλοί άλλοι και το ε, παρατηρητήριο επιχειρήσεων επίσης, το οποίο βέβαια φαίνεται πως ετάσσεται υπέρ των πολυεθνικών κολοσσών η τεχνολογία, οι, επιχειρη... οι τεχνολογικές ε, βέβαια επιχειρήσεις νομίζω πως έχει καταστεί σαφές ότι προσπαθούν να αποδυναμώσουν τον... το κείμενο και να γίνουν την πλάστιγκα υπέρ τους. Ο κύριος ε, Φως επίσης ασχολήθηκε υπέρ το δέον με τα μέσα ενημέρωσης, ε, με τον τύπο και όχι με ε, τις επιχειρήσεις τεχνολογίας. Και φυσικά δεν είναι μυστικό το γιατί. Τώρα, όταν κάποιος ε, έχει ένα κείμενο τεσσάρων σελίδων, δεν νομίζω πώς μπορεί να μιλήσει περί διαφάνειας. Αντιθέτως, μας λέτε. Αυτά, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε εδώ τη δική μου θέση. Δίνω μάχη γι' αυτό εδώ και 15 χρόνια περίπου και αυτό μου επέτρεψε να εργαστώ σκληρά ε, για το κείμενο αυτό όταν επιτέλους η Κομισιόν μας πρότεινε κάτι κάπως ουσιαστικό. Το κείμενο λοιπόν που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Είχα ζητήσει να παρέμβω πρώτος όμως καθώς ο κύριος Βόμποντα μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω ε, στην Προεδρία αποφάσισα να μην παρέμβω πρώτος, να αφήσω τη δυνατότητα στον καθένα να, να πάρει το λόγο. Εδώ και πολλά χρόνια αναρωτιέμαι το εξής. Και είναι σοβαρό το ερώτημα αυτό. Εάν αντί να μιλάμε για δωρεάν ίντερνετ, ελεύθερο ίντερνετ, μιλούσαμε για κάποιο αγαθό, για κάποιο εμπόρευμα, θα ήταν πολλοί αυτοί εδώ που θα θεωρούσαν ότι τα εμπορεύματα αυτά τα οποία παράγουν κάποιοι εργαζόμενοι σε επιχείρησεις που θα ήταν υπέρ αυτά τα εμπορεύματα να είναι δωρεάν, να είναι ελεύθερα στην πρόσβαση, να μπορεί κάποιος να πηγαίνει όπως στα μαγαζιά, όπως το, στις του Amazon και να παίρνει στην αποθήκη του Amazon ό,τι θέλει, χωρίς να πληρώνει τίποτα. Φυσικά και όχι. Θα θέλαμε αυτό να το οργανώσουμε. Είναι, έχουμε παραγωγή, έχουμε μισθούς, έχουμε κατανάλωση. Πώς λοιπόν ε, υπάρχει αυτή η υποταγή εδώ και κάποια χρόνια και δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό από ένα αυτοκίνητο ή από γλυκά ή από ένα ρούχο ή από ένα απλό εμπόρευμα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η προπαγάνδα ε, και έχει δίκιο κύριε για να θυμώνει που μας έχει οδηγήσει ε, στο να μην θέλουμε ε, να έτσι να δώσουμε μια σκηνή εικόνα στους νέους τόσο εισαγωγικών ή σε κάποιους νέους δεν είναι όλοι νέοι έτσι το, η κάθε εργασία θα πρέπει να πληρώνεται εκτός εκτός από ό,τι φαίνεται να ακούσω κάποιους που μου εδώ αυτοί, αυτοί που δεν φτιάχνουν πράγματα με υφάσματα και με ε, εργαλεία απλά γράφουν με ένα στυλό ή δουλεύουν σαν υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει πλέον οικονομία για τους καλλιτέχνες, δεν θα υπάρχουν πια καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες πρέπει να μπορούν να φάνε, να ζήσουν, να θρέψουν την οικογένειά τους. Δεν μπορούμε να τους πούμε να πάνε στο εργοστάσιο όλη μέρα και το βράδυ να παίξουν και λίγη μουσικούλα. Δεν είναι έτσι. Εγώ κοίταζα τα αριθμητικά στοιχεία. Εδώ και, κά, πέντε χρόνια ούτε μία από τις γκάφα, των οποίων τα κέρδη δεν αυξάνονται. Έτος με το έτος. Το ταλέντο λοιπόν ε, και ακούσαμε πολλά τέτοια και εδώ και αλλού Βεβαίως και είναι ε, σεβαστό. Δεν θα κλάψουμε γι' αυτό όμως. Μιλάμε για καπιταλιστές που χρησιμοποιούν την προπαγάνδα για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν πώς η Ευρώπη, η οποία ήταν εξαιρετική στον γενικό κανονισμό προσωπικών δεδομένων, δεν μπορεί να είναι τόσο εξαιρετική για τα συλλογικά δεδομένα. Και στα συλλογικά αυτά δεδομένα βεβαίως υπάρχουν τα ωράρια, τα ξενοδοχεία όπου κλείνουμε, έγινε σχετική αναφορά νωρίτερα. όμω υπάρχουν και πολύ πιο πολύτιμα πράγματα. Ο τύπος, ο τύπος θα εκλείψει. Α δώσουμε πληροφορία, το έχω ξαναπεί νομίζω πριν από μερικού μήνε. Στη Γαλλία έχουμε διαπιστώσει από τον, τον Ιανουάριο τον Αύγουστο του 2018 7% των κερδών έφυγε από τον τύπο και πήγε προς το ψηφιακό, ψηφιακό τομέα επί 10 χρόνια ή και επί 5 χρόνια μας συνεχιστεί αυτό, δεν θα αντέξει ο τύπος. Οπότε, αν θέλετε να πεθάνει ο τύπος, ψηφίστε αυτά που σας λέει η γκάφα να ψηφίσετε. Να πω ακόμα παραπέρα. Η δημιουργία, η καλλιτεχνική, δεν είναι αυτό που κάνουμε όταν τελειώσουμε τη δουλειά μας. Ή επειδή, ξέρω εγώ, ε, είμαστε συνοχωρημένοι και δύο μέρες που έχουμε άδεια θα γράψουμε ένα τραγούδι. Όχι είναι κάτι στο οποίο δεσμεύεται ένας καλλιτέχνης. Θέλετε να μην ζει από αυτό, το δέχεστε αυτό, να πεθαίνουν τη πείνας. Ποιοι είμαστε εμεί για να μπορούμε να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Βέβαια υπάρχουν οι νέοι, του έχουμε συνηθίσει. Έχετε δίκιο, κύριε Άντερσον. Ε, ναι, κύριε Ρέρα, του έχουμε συνηθίσει. Ο ρόλο μα ω δημόσιοι παράγοντε, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, θα έπρεπε να είναι να του εκπαιδεύσουμε να, για να καταλάβουν ότι κάθε αντικείμενο, κάθε ιδέα, κάθε καλλιτεχνικό έργο πρέπει κάποιος να το πληρώνει. Και το καλό είναι ότι δεν πληρώνουν αυτοί. Δεν ζητούμε από να το πληρώσουν, ζητούμε από επιχειρήσει να το πληρώσουν. Από τι γκάφα. Νομίζω ότι από ηθική πλευρά η άποψή μα είναι εξαιρετική, δεν βλέπω γιατί δεν υπερασπιζόμαστε. Βεβαίω υπάρχουν προβλήματα με τα φίλτρα. Δεν υπάρχουν όμω φίλτρα έχει αποσυρθεί αυτό. Κάποιοι θα πούν, και εγώ μάλιστα δίσταζα, ε, ότι υπάρχει ανάγκη να πούμε αν ένα προϊόν είναι ελεύθερο ή όχι. Σα βλέπω ότι χαμογελάτε κυρία Ρέντα. Αν όμω ε, πάω να πάρω το παλτό σα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, είναι δικό σα το παλτό. Εσεί όμω, η μεν και η δε που σα άκουσα προηγουμένω, προσπαθείτε, ναι, ναι, ναι, γελάστε, θα δείτε μετά τι επιπτώσει. Εγώ δεν γελούσα όταν μιλούσατε, έτσι. Δεν υπήρχε και λόγο να γελάσω βέβαια. Γελάστε λοιπόν. Δίνετε όμως το χέρι εδώ και βοηθάτε σε μια τεράστιο εγχείρημα αρπαγής περιεχομένου. Δεν και δεν γίνεται δωρεάν αυτό που λέτε. Υπάρχουν κέρδη. Και ποιο τα παίρνει τα κέρδη αυτά. Τα, παίρνει, ε, τα παίρνουν οι δημιουργοί ή ο τύπος. Ο τύπος είναι η πιο στέρεα βάση για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία, δικαστική εξουσία, ανεξάρτητη και ανεξάρτητη, ανεξάρτητος τύπος. Τι γίνεται, ε, λοιπόν, ποιοι γράφουν τώρα στη Μοντ, παραδείγματος χάρη, το YouTube, το Google, καλά, καλά νέα, κακά νέα, ψευδή νέα, φήμες, βία και από αυτά βγάζουν, βγαίνουν χρήματα. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε μια κάποια ηθική προσέγγιση για το θέμα αυτό. Ποιοι είμαστε εμεί οι Ευρωπαίοι που θέλουμε να φτιάξουμε ε, μια κοινωνία που θα ζούμε όλοι μαζί και θέλουμε να φτάσουμε σε συγκεκριμένο επίπεδο πολιτισμού. Θα τα αποφασίζουν αυτό κάποια αλγόριθμοι. Κανεί δεν θα άφηνε στα, στα δίκτυα να μπουν τέτοια πράγματα στα δικά του. Ενώ τα κάνουν αυτοί. Παιδική πορνογραφία, ε, άρνηση ολοκαυτώματο και ό,τι άλλο θέλετε. Το κείμενο λοιπόν αυτό δεν είναι τέλειο. Κανένα κείμενο μας δεν είναι τέλειο. Από ανθρώπου ε, εκπονούνται αυτά. Εδώ και 15 χρόνια που είμαι εδώ όμως, ποτέ δεν έχω δει τόση βία κατά ενός νομοθετικού οργάνου. Όχι μόνο μάλιστα ενό νομοθετικού οργάνου, κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί έχουν διεισδύσει στο Συμβούλιο. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ να πιστέψω ότι ένα μέρος των κρατών που είναι κατά δεν έχουν τράπεζες όπου καταθέτουν τα χρήματα τους η γκάφα. Και με προκαλείται γιατί μπορώ να δώσω και στοιχεία. Θα τα αφήσουμε να περάσει αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο καθένα θα λάβει τι ευθύνε του, βεβαίω. Και βεβαίω ε, ο ψήφο του καθενό είναι σεβαστή. Είναι όμω φοβερό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρομερό αυτή η προπαγάνδα έχει διεισδύσει και στα τρία θεσμικά οργανωτικά, κάτι που δεν έχω δει εγώ ποτέ, ακόμα και στον διαθεσμικό διάλογο. Είναι σαν η Google να είναι στο Συμβούλιο ε, Υπουργών της Σουηδίας και να λέει, ξέρετε, αυτή τη φορολογική, ε, ε, το φορολογικό μέτρο εγώ δεν το θέλω. Δεν ήταν η Google, ήταν η YouTube όμως, στο Στρασβούργο, το Δεκέμβριο. Πώ μπορούμε να δεχτούμε εμεί κάτι τέτοιο, εμεί που αναπτύξαμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την οποία μα ζηλεύουν οι Αμερικανοί. Λέω λοιπόν ότι το κείμενο αυτό είναι ακονοποιητικό, είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα για να δώσουμε ένα δικαίωμα ε, στους δημιουργούς, να δώσουμε κάποια δικαιώματα. Δεν πρόκειται λοιπόν να υπογραμμίσω αυτά που είναι καλά, τα είπε ο εισηγητής, τα είπαν και άλλοι. Είναι όμως πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα. Κάποιοι από εμά ετοιμάζονται να δώσουν χέρι σε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επιζήμιο και θα μας κρίνει η ιστορία γι' αυτό και που έχει σχέση αυτό με τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο που το σκεφτόμαστε και το συζητάμε εμεί εδώ οι Ευρωπαίοι και όχι οι Αμερικανοί ή ότι οι Κινέζοι δεν του νοιάζει καθόλου. Είναι επειδή αυτό που εμεί ζητούμε σε επίπεδο ελευθερία θα διαλυθεί από μια προπαγάνδα, από ένα καπιταλισμό και από τη δημιουργία ιδεών που είναι στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων στην πολιτεία στο Κογκρέσο, γίνεται συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να διαλυθεί το Google και εμεί θέλουμε εδώ ε, να το ενισχύσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλετε το λόγο, κύριε Άντερσον, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ, κύριε Φως, που μου είπατε να ανοίξω το μικρόφωνο. Το θυμήσατε. Δεν θα έπρεπε να είχα γελάσει όταν μιλούσε ο πρόεδρος. Όλα θυμάμαι... δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά θυμάμαι λοιπόν την ιστοσελίδα του. Όχι, όχι κύριε πρόεδρε, ε, εγώ δεν έδειξα σωστή συμπεριφορά. Θυμάμαι λοιπόν ε, πριν ε, επιβληθεί στη Γαλλία η ελευθερία της ε, φωτογραφίας και υπήρχε μια φωτογραφία στο site του Κοινοβουλίου η οποία αποτελούσε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ο πρόεδρος ο, ο οποίος ο ίδιος παραβίασε την νομοθεσία μας λέει τα αντίθετα μας λέει ότι ε, θα πρέπει να απαγορεύεται το ανέβασμα περιεχομένου, να απαγορεύεται να, ε, ανεβάζουμε συνδέσμους ε, σε άλλες, για άλλες σελίδες. Απαγορεύονται διάφορα πράγματα που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα, όμως υπάρχει φίλτρο και επιβάλλεται φιλτράρισμα αυτόματο από αλγορίθμους. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι το ίδιο αυτό με το να πάρετε το παλιτό που ανήκει σε κάποιον άλλο. Και στην ουσία εδώ δημιουργείται περισσότερη σύγχυση παρά σαφήνεια. Βέβαια, σίγουρα θα έπρεπε να μην γελάσω και να μείνω απρόσωπος γιατί τέτοιος πρέπει να είναι ο πολιτικός. Ένα ερώτημα Είπατε ότι υπάρχει μια φωτογραφία στην ιστοσελίδα μου που δεν έχει τα δικαιώμα, το δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Ή δεν κατάλαβα καλά. Yes, you, you have website committed. Ναι, ναι, στο, στον ιστοτοπό σα. Ναι, ναι, παραβιάστε δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Είναι ελεύθερη φωτογραφία που μου έδωσε το δικαίωμα το κοινοβούλιο να σε Δεν υπάρχει νομίζω κάτι τέτοιο θέμα. Σα ευχαριστώ πολύ ο εισηγητής. Λοιπόν, καταρχά σας ευχαριστώ για αυτήν την ε, πλούσια, πλουσιότατη ανταλλαγή απόψεων η οποία βέβαια πήρε λίγο διαφορετική τροπή, προσπάθησε ο ένας να απαξιώσει τον άλλον. Βέβαια το θέμα εδώ είναι να υπάρξει ένας προσανατολισμός και να εξετάσουμε το ερώτημα του τι μας περιμένει. Τέλος πάντων, τέλος πάντων θα προσπαθήσω να ε, εστιάσω κι εγώ πρώτα Ρωτήθηκα αν θα καταφέρουμε σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο να ε, μεταφέρουμε την ε, έννοια του ε, δημιουργού, της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά και θα πρέπει να μας απασχολήσει, όμως βέβαια σε συνδυασμό με αυτό θα πρέπει να κάνουμε και το ερώτημα του του συνδυασμού αυτού με τον σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων. Τώρα, δεν ε, τέθη ποτέ το ερώτημα το πόσο ε, ποιος ε, θα πρέπει να δημοσιευτεί ποιος θα έχει τα δικαιώματα, οι πλατφόρμες, ο δημιουργός κτλ. Όχι. Ε, τα δικαιώμα, ε, το που πρέπει να ισχύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν συζητήθηκε ποτέ, δεν ετέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα. Εμείς προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ε, του δημιουργού. Όμως πρέπει να εξετάσουμε και τις συνέπειες ενός ψηφιοποιημένου κόσμου. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Επίσης, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα μόνο ε, θεμελιώδες δικαίωμα, δηλαδή της ελευθερίας έκφρασης, αλλά θα πρέπει αυτό να συνεπάρχει και με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Και εδώ δημιουργούνται οι προστριβές, οι διαφωνίες, ε, εδώ υπάρχουν ε, παρεξηγήσεις, ο ένας λέει δεν με σέβεστε κτλ. Όμως έχουμε δύο θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία αμφότερα πρέπει να αποτελούν ε, βάση, θεμέλιο και μέτρο σύγκρισης ταυτόχρονα. Βέβαια, μου ασκείται κριτική για το ότι η διαδικασία έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Θα απαντήσω ότι όχι και μάλιστα εσείς δεν συμμετείχατε στη διαδικασία για να ε, το ξέρετε. 13 ε, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε, καταχύμωνο τελειώσαμε, μήνες κράτησε η δουλειά και η τελική ε, ψηφοφορία προβλέπεται για τις 18 ε, Απριλίου. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να ολοκληρώσουμε, διότι αυτό είναι και απόδειξη της δικής μας πολιτικής βούλησης. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάποια πράγματα, να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για να μην χρονοτριβούμε και να μην τραβήξουν εσαΐ. Δεν γίνεται λοιπόν να έχουμε φτάσει στο τέλος τη κοινοβουλευτική θητεία, να έχουμε φτάσει τόσο μακριά στον τριμερή διάλογο και να μην ψηφίσουμε. Ελπίζω λοιπόν να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα, ως ε, προς το κείμενο, καταλαβαίνω βέβαια ότι όσοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία έχουν ε, ερωτήσεις ε, για το κείμενο. Βέβαια να σας πω ότι πρόκειται για μια ανεπίσημη εκδοχή του κειμένου. Αυτή τη στιγμή η γραμματεία εργάζεται πυρετοδός μαζί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα έτσι ώστε να ε, συνταχθεί μια ε, επίσημη εκδοχή. Όμως εφόσον το επιθυμείτε μπορούμε να σας ε, δώσουμε την, το ανεπίσημο κείμενο. Τώρα, όσοι ακολούθησαν βήμα-βήμα τη διαδικασία και παρόλα αυτά κάνουν τέτοια σχόλια, ε, δεν είστε σοβαροί. Τώρα, ως προς το περιεχόμενο, εδώ εντάξει, φτάσαμε στα άκρα. Τώρα, λέτε ότι στους ορισμούς υπάρχει εξαίρεση για τις ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ναι, εντάξει. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει και μία νέα διάταξη για ε, τεστ ε, αναλογικότητας. Όταν, ας πούμε, μία πλατφόρμα δεν έχει ας πούμε μέχρι 5 εκατομμύρια χρήστες, ε, μέχρι 5 εκατομμύρια ε, θεάσεις το μήνα, αλλά 5 εκατομμύρια 0,0001. Εντάξει, δεν θα, το, δεν θα τη βάλουμε στο ίδιο καζάνι με τους ε, κολοσσούς. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει κάποια αναλογικότητα. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο. Υπάρχουν εξαιρέσεις που προβλέπονται. Και α είμαστε λογικοί. Τώρα, η κυρία Κάουφμαν με ρώτησε τι συμβαίνει με αυτές τις εξαιρέσει και πώς καταλήξαμε εκεί. Στη διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου υπήρχε μία εξαίρεση για επιχειρήσεις με ε, κύκλο εργασιών μέχρι 10 ε, εκατομμύρια το χρόνο. Ε, εκεί ακριβώς ήταν το σημείο στο οποίο έγιναν οι συγκρούσεις ε, με το Συμβούλιο και ψάξαμε να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Το ένα κράτος ε, μέλος ήθελε να συμπεριληφθεί αυτή η διέταξη στο άρθρο 13. Ένα, ένα άλλο κράτος μέλος ήθελε διαφορετική ειδική μεταχείριση για τους ε, νέους, για τις νέες επιχειρήσεις και καταλήξαμε να συμφωνήσουμε σε κάποια κριτήρια. Αυτά τα 10 εκατομμύρια δηλαδή δεν ε, ήταν ουρανοκατέβατα. Υπήρχε μια βάση από την Κομισιόν πάνω στην οποία στηριχθήκαμε. Και καταφέραμε λοιπόν να βρούμε έτσι μια ικανοποιητική τάξη μεγέθους και ε, για όλους έτσι ώστε οι πολύ μικρές πλατφόρμες να μην κληθούν να ε, επομιστούν τεράστιο κόστος και να μην πληρώσουν τα σπασμένα. Τώρα φτάσαμε βέβαια και στην αξιολόγηση. Και ακριβώς επειδή υπήρχαν οι διαφωνίες στο Συμβούλιο και κράτησαν βδομάδες, μας κόστησαν πολύ χρόνο, καταλήξαμε στο ότι υπήρξε αυτό το μπλοκάρισμα. Δεν βρήκαμε πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, οι ισορροπίες ήταν λεπτές, ε, κόλλησε το θέμα για πολύ καιρό και έπρεπε να γίνουν αμοιβέ υποχωρήσει. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθήσαμε στη νομική δομή να πάρουμε τους ορισμούς και να ε, συγκρίνουμε τι έγινε και με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γι' αυτό και έγινε ότι έγινε με το άρθρο 13, διότι η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει και τις ε, λεγόμενες παθητικές πλατφόρμες, τις μη ενεργές πλατφόρμες. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να περιορίσουμε κάπως το φάσμα έτσι ώστε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα και των μικρότερων επιχειρήσεων. Γι' αυτό προέκυψαν εξαιρέσεις. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω αυτή την κριτική που ασκήθηκε, που λέτε ότι τα τραβήξατε στα άκρα όλα. Προσπαθήσαμε να τηρήσουμε την αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, τα φίλτρα, τα αυτόματα φίλτρα για το ανέβασμα περιεχομένου δεν υπάρχουν στο κείμενο. Εδώ βέβαια το πρόβλημα είναι στην πράξη, όταν δηλαδή υπάρχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με, τον, με, το οποίο ο χρήστης ανεβάζει ό,τι θέλει, αλλά ο χρήστης δεν αποφασίζει και δεν μπορεί να κρίνει τι είναι, προστατεύεται, από, τι έχει δικαιώματα και τι όχι, θα πρέπει την ευθύνη να φέρει η πλατφόρμα στην οποία ανεβαίνει αυτό το περιεχόμενο. Και σε αυτήν την περίπτωση, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να κρατήσουμε υπόλογους όλους τους ε, χρήστες που ανεβάζουν το περιεχόμενο, να ε, έχει την ευθύνη η πλατφόρμα για να κάνει αυτή τη διαλογή. Γι' αυτό νομίζω είναι απόλυτα αιτιολογημένο ε, το σκεπτικό του να φέρει η πλατφόρμα την ευθύνη, διότι αυτή στην ουσία κερδίζει χρήματα και αυτή λοιπόν θα πρέπει να διαχειρίζεται τις ε, άδειες. Και το θεωρώ λοιπόν απόλυτα αιτιολογημένο. Η διαχείριση της ευθύνης λοιπόν είναι αρμοδιότητα της πλατφόρμας, διότι η πλατφόρμα έχει ευθύνες, έχει και κέρδος. Όταν, ας πούμε, ανοίγω ένα εστιατόριο, δεν μπορώ να πω, ναι, είμαι πάρα πολύ μικρή επιχείρηση, γι' αυτό, λοιπόν, δεν χρειάζεται να τηρήσω ε, τις, ε, τα πρότυπα, τα υγειονομικά πρότυπα. Πρέπει να προσαρμοστεί το επιχειρηματικό μοντέλο, διότι θα πρέπει πέρα από την ευθύνη της ε, υποδομής να υπάρχει και ευθύνη ακριβώ διότι οι πλατφόρμες αυτές έχουν κέρδος. Και νομίζω πως είναι προφανές λοιπόν γιατί ε, υπάρχουν αυτές οι εξαιρέσεις στο άρθρο 13. Τώρα αυτές οι επιγραμμικές πλατφόρμες γνωριμίων νομίζω είναι αυτονόητο γιατί εξαιρούνται. όταν κάποιο ανεβάζει μια φωτογραφία του, είναι ο ίδιος κάτοχος των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Εννοείται λοιπόν ότι δίνει τη συγκατάθεσή του όταν ανεβάζει ο ίδιος μια φωτογραφία του εκεί πέρα. Βλακίες λοιπόν είναι αυτά που ακούω ότι είναι, ας πούμε, δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πλατφόρμες γιατί κάποιο ε, θέλει να στερήσει δικαιώματα κτλ. Τώρα άρθρο 11. Στο άρθρο 11 αναφέρεται ρητά η συμμετοχή των δημοσιογράφων. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός ανάμεσα σε ελεύθερους επαγγελματίες ή σε ε, που εργάζονται με σύμβαση σε οτιδήποτε άλλο. Ίσως έγινε παρερμηνία ε, διότι ακριβώς στην ε, στρατηγική σκέψη δεν αναφέρεται ότι το κράτος μέλος θα πρέπει να διεξάγει τους ε, κατάλληλους ελέγχους, έτσι ώστε να αποφεύγονται τέτοιες περιπτώσεις. Για μένα αυτό είναι παρερμηνία. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει τώρα αυτό δεν ε, τους επηρεάζει όλους, το 11-5 νομίζω, νομίζω σε αυτή την παράγραφο αναφέρεστε. Θα το ψάξω βέβαια. Όμως αναφέρεται ρητά ότι όλοι οι δημοσιογράφοι συμμετέχουν. Δεν γίνεται κανένας διαχωρισμός ανάμεσα σε υπαλλήλου και ελεύθερους επαγγελματίε. Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική χρήση τώρα. Ο πολίτης μπορεί να χρησιμοποιεί αποσπάσματα από άρθρα για προσωπική του χρήση, να τα ανεβάσει δηλαδή σε μια πλατφόρμα. Η πλατφόρμα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένη να ζητήσει άδεια διότι πρόκειται για μία ενέργεια, για ανέβασμα περιεχομένου το οποίο έχει λάβει έγκριση. Είναι δηλαδή για ιδιωτικού σκοπού. Ο χρήστη λοιπόν μπορεί να ανεβάσει κάτι για προσωπική χρήση. Τώρα, αν μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει περιεχόμενο που έχει ανέβει, ένα άρθρο ας πούμε για προσωπική του χρήση, αυτό είναι μία άλλη ερώτηση, είναι λίγο πιο λεπτό το ζήτημα. Ή αν κάποιος ανεβάσει έναν σύνδεσμο που οδηγεί σε έναν οργανισμό μέσων ενημέρωσης και αυτό θα πρέπει να το ε, δούμε. Όταν πρόκειται όμως για προσωπική χρήση, αυτό επιτρέπεται. Τι άλλο. Α, ναι. Πλήρης εναρμόνιση ή όχι. Ναι, είχε γίνει μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Από τη μία, τα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας είναι πλήρως, εντελώς κατακαιρματισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια κρατημέλη έχουν ε, πιο ε, συνολική νομοθεσία, κάποια όχι, κάποια, σε κάποια κράτη-μέλη είναι τελείως άγνωστη αυτή η έννοια. Υπάρχουν λοιπόν τεράστιες διαφορές. Γι' αυτό προβλέπεται μία εξαίρεση για καρικατούρα, για σάτυρα, για έτσι, διάφορα αποφθέγματα, παροδίες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργούνται προβλήματα σε τέτοιες ε, περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο και οριακό να καθοριστεί ο τύπος της χρήσης ενός ε, περιεχομένου. Όμως αναφέρουμε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις, παρόμοιες ε, δομές, τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επικεντρώνονται στο τέλος, στον στόχο και αυτό να προσπαθούν να τηρείται. Δεν προσπαθούμε δηλαδή με την οδηγία να φτάσουμε σε πλήρη εναρμόνιση. Ωραία θα ήταν, βέβαια, να υπάρχει ένας ε, κανονισμός ε, για το ψηφιακό περιβάλλον που να παρέχει πλήρη εναρμόνιση. Όμως εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορές. Το καθένα είναι περήφανο για τον τρόπο που χειρίζεται αυτά τα θέματα και εδώ δεν μπορούμε να παρέμβουμε και πολύ. Τώρα, οι εξαιρεσει ε, που προέρχονται από πιέσεις ε, λόμπι. Τώρα, όταν κατηγορείται ένας ε, συνάδελφος για το ότι έχει δεχτεί πίεση από λόμπι και για... επειδή εκφράζει την προσωπική του άποψη, αυτό για μένα είναι άστοχο πρέπει να έχουμε το δικαίωμα τη άποψή μα και να λέμε πούμε, ότι για παράδειγμα για τις ε, επιγραμμικέ πλατφόρμες ε, γνωριμιών εμείς ε, θέλουμε εξαίρεση. Οι εξαιρέσει που έχουν προκύψει έχουν προκύψει για κάποιους λόγους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για παράδειγμα, όταν κάποιος έχει μια πλατφόρμα, θέλει να ανεβάσει κάτι, και οι λεπτομέρειες δεν ε, εμπίπτουν στη, στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 13, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να το κάνει. Θα πρέπει δηλαδή ας πούμε, να υπάρχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση κτλ. Στις περιπτώσεις αυτές όμως, στις ε, επιγραμμικές πλατφόρμες γνωριμιών, αυτό δεν είναι εφικτό, διότι είναι αντίθετο στο σκοπό ύπαρξης αυτής της πλατφόρμας. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε τι πραγματικά θέλουμε και γι' αυτό καταλήξαμε στον ορισμό που καταλήξαμε. Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα σκέψης και όχι πίεσης από λόμπι. Είναι λοιπόν απόφαση κατόπιν όριμης κριτικής σκέψης και δεν μας είπε κανείς τι θα κάνουμε. Επειδή λοιπόν ακριβώς δεν υπάρχει τέτοια αναφορά στον ορισμό, συμπεριλάβαμε και έναν αρνητικό κατάλογο, έτσι ώστε να παρέχονται αναγκαίες διευκρινήσεις. Τώρα η κυρία Χάουταλα αναφέρθηκε σε, στο, σε κάποια πράγματα ότι ποιος μίλησε με ποιον, ποιος δεν ζήτησε τη γνώμη ποιου. Υπάρχει και το δικαίωμα πρωτοβουλίας, ξέρετε. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω με όλους, να ακούσω την άποψη όλων των πλευρών. Τώρα αν ξέχασα κανέναν, δεν ξέρω, ελπίζω πως όχι, αλλά γιατί δεν ήρθε να με βρει κάποιος αν θεωρούσε ότι χρειάζεται. Τώρα, άρθρο 13. Δείτε τη δομή. Αναφέρεται σε ενεργές πλατφόρμες οι οποίες φιλοξενούν περιεχόμενο που ε, έχει δικαιώματα. Προστατεύεται από δικαιώματα. Εάν αυτό συμπεριέλαβε και τις ε, νεοφύσεις επιχειρήσεις, τότε θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει να περιέχεται και στο άρθρο 2, παράγραφος 5. Τώρα, προσπάθησα να δώσω όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να εξαντλήσω τη συζήτηση για όλα τα θέματα. Ελπίζω να απάντησα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις ε, ε, πληροφορίες και τώρα θα ακούσουμε πώς θα συνεχιστεί. Η κοινή ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 15.45 ε, θα ψηφίσουμε δηλαδή για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το, περιεχόμενο, το ψηφιακό περιεχόμενο. Έκτακτη συνεδρίαση 26 Φεβρουαρίου ε, τρίτη στις 3 το μεσημέρι και επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 3. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για την ε, ε, συμμετοχή σας στη σημερινή συζήτηση και να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς που σήμερα είχαν κάπως πιο δύσκολη δουλειά από ό,τι συνήθως γιατί είναι πολύ τεχνικά τα θέματα. Σας ευχαριστώ όλους.